Hello time to... Καλώς ορίσατε όλοι. Ήρθε η ώρα να αρχίσει η συνεδρία αυτή τη Επιτροπής. Καλώς ορίσατε όλοι. Περνάμε στο πρώτο μέρος ε, της ημερήσιας διάταξης, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη. Βεβαίω, πολύ ωραία, ευχαριστώ. Περνάμε στο δεύτερο μέρος, οι ανακοινώσει της Προέδρου. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχετε ήδη ενημερωθεί ότι ε, η ανακοίνωση των υποψηφίων του ε, βραβείου Σαχάροφ για το 2018 θα γίνει την 5η 27 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στην αίθουσα Jan 2Q2 μαζί με την Επιτροπή ΑΦΕΤ και την η, την υποεπιτροπή ΔΡΟΑ. Η Λίντα Μακέβαν δεν θα μπορέσει να παραστεί λόγω άλλων υποχρεώσεων της εκτός Βρυξελών. Όμως θα παρευρεθώ εγώ ως συμπρόεδρος εκ μέρους της. Ελπίζω ότι, ότι θα εκπροσωπηθεί πολύ ωραία και η Επιτροπή μας. Περνάμε στο τρίτο σημείο. Η έγκριση των αποφάσεων και συστάσεων των συντονιστών. Οι αποφάσεις και συστάσεις των ε, συντονιστών μετά τις συνεδρίες της 29ης Αυγούστου φέτος ε, βρίσκονται στους ε, φακέλους σας. αν δεν γίνουν παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί. Έχετε τον κατάλογο, τον οποίο παρακαλώ να ελέγξετε δηλαδή. Κατόπιν το επόμενο θέμα είναι οι ανακοινώσεις της Επιτροπής. Το σημείο αυτό των ανακοινώσεων της Επιτροπής είναι μόνιμο θέμα στην ημερήσια διάταξη και νομίζω ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Θα ήταν καλύτερα αν η Κομισιόν συνηθίσει να μας ενημερώνει παραδείγματο χάρη για τις ανακοινώσεις τις οποίες προετοιμάζει. Πριν από δύο εβδομάδες η Επιτροπή δημοσίευσε μία ανακοίνωση για πιο αποδοτική ε, αρχιτεκτονική, ε, χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για τις επενδύσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια άλλη για τη νέα συμμαχία Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας. Μήπως μπορείτε να μας πείτε σε ποια κείμενα ε, ποια κείμενα επεξεργάζεστε αυτή τη στιγμή και μήπως μπορούμε να ε, συμφωνήσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το θέμα των ανακοινώσεων για το σκοπό αυτό στις επόμενες συνεδριάσεις μας. Θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους της Επιτροπής, στον Κάρστεν Σόρενσεν. Θέλετε να πείτε δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, που μας δίνετε να την ευκαιρία να μιλήσουμε. Ε, σημείωσα τα όσα είπατε και σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρησή σας. Πράγματι αναφερθήκατε σε δύο σημαντικές ανακοινώσεις επί των οποίων θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας. Και φυσικά είμαστε ιδιαίτερος ευτυχείς να εκπροσωπούμαστε στο κατάλληλο επίπεδο στην Επιτροπή σας για να σας ενημερώνουμε για όπως πιστεύετε ότι πρέπει για τα δύο αυτά θέματα. Ένα τρίτο που θέλω να αναφέρω είναι η ανακοίνωση που ονομάζεται «Διασυνδεσιμότητα Ασίας, Asia Connectivity και έχει πλήρη τίτλο Σύνδεση Ευρώπης-Ασίας ε, οικοδόμηση μιας πλήρους στρατηγικής. Και επίσης μπορούμε να σας ενημερώσουμε όπως επιθυμείτε. Και, εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω ότι αυτά τα οποία είπατε τα σημειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την απάντηση, λέει η Πρόεδρος. Χαίρομαι που μαθαίνουμε τα, τις εξελίξεις. Υπάρχουν ε, ερωτήσεις επ' αυτού. Αν όχι, περνάμε στην ακρόαση. Το πρώτο θέμα μας αφορά την ακρόαση με θέμα την συμμετοχή της ε, Αφρικανικής Διασποράς στην Ευρώπη για την πρόθεση των αποτελεσματικών αναπτυξιακών πολιτικών συνεργασίας. Οπότε απευθείας πλέον θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους την Σεσίλ Κέγκε, τη Σεσίλ Κασέτου Κέγκε, η οποία είναι η συντονίστρια. Χαίρομαι πολύ που βρίσκεσαι εδώ. Και έχουμε επαρκή χρόνο για να συζητήσουμε και να ακούσουμε απόψεις επί του θέματος. να Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι Μύρια που μου δίνετε το λόγο και την Προεδρία αυτής της ε, δημόσιας ακρόασης. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους, αγαπητοί προσκεκλημένοι, συνάδελφοι, ε, ακροατήριο. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ε, ε, για την συμμετοχή σας στην ακρόαση. Έχουμε προθεσμία μέχρι τις 5 παρατέταρτο, οπότε επαρκεί χρόνο για συζήτηση. Όμως τότε προβλέπεται ψηφοφορία, οπότε πρέπει να σταματήσουμε για να γίνει ψηφοφορία. Έχουμε καλέσει τέσσερις ομιλητές, πιο συγκεκριμένα δύο ε, ομιλήτριες και δύο ομιλητές, τους οποίους θα σας παρουσιάσω εντός ολίγου. Ε, έχουν συνολικά περίπου 30 λεπτά, ο καθένας για την ε, αρχική του παρέμβαση. Θα ακολουθήσει μια ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές. Οπότε, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θέλω να σας παρουσιάσω τους τέσσερις ομιλητές. Καταρχήν, η κυρία Μαρίνα Μάνκε, την οποία βλέπετε εδώ εκ δεξιών μου, επικεφαλής ε, του τμήματος ε, επαγγελματικής κινητικότητας ε, και ανθρώπινης ανάπτυξης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και θα μας μιλήσει για την, το ρόλο της Διασποράς ως εταίρου για την ανάπτυξη της εφαρμογής του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη Μετανάστευση. Επίσης θα μας δώσει μια περιγραφή των τάσεων, των στοιχείων και επίσης τα μαθήματα που έχουμε μάθει από την Διασπορά της Αφρικής. Εκ μέρους της Αφρικανικής Διασπορά, Διασποράς των Βρυξελών θα μας παρουσιάσουν την, ε, τα θέματα της Αφρικανικής Διασπορά, Διασποράς στην Ευρώπη, όπως επίσης και κάποιες πρωτοβουλίες της Αφρικανικής Διασποράς. Οι ομιλητές είναι η Μαρί Σοντάλ Ουιτόνζε, ιδρύτρια και πρόεδρος της ADNE, που είναι το δίκτυο της Αφρικανικής Διασποράς στην Ευρώπη, με έδρα της Βρυξέλλης, και ο κύριος Τιαρνός Αιντού που είναι σύμβουλος των Σούμαν Associates, Associates επίσης της Βρυξέλλης, εξ αριστερών μου. Η πρώτη, η κυρία Ουιτόνζε, θα μας εξηγήσει πώς το δίκτυο ενθαρρύνει την μεγαλύτερη συμμετοχή Αφρικανών ανδρών και γυναικών στην οικοδόμηση Αφρικής και θέλει να βοηθήσει με τη δημιουργία πλατφόρμας και διαβουλεύσεων ανταλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Διασφοράς. Ως βασικός παράγων της ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη σε, που αφορά μια σειρά σημαντικά θέματα ε, στον τομέα της πολιτικής, τα θεσμικά θέματα, αλλά επίσης ε, και τον πολιτιστικό τομέα. Ο κύριος Διόπ θα ασχοληθεί περισσότερο με την οικονομική πτυχή και την συνεισφορά της διασποράς στην ανάπτυξη Αφρικής συγκεκριμένα τις ιδιωτικές επενδύσεις. Πιθανόν αναφερθεί και στο ρόλο της διασποράς στον βασικό τομέα της ε, εκπαίδευσης υγείας στην Αφρική. Τέλος, ο κύριος Hans Stausboll, ε, ελπίζω να μην σκόντωσα το όνομά σου, είναι διευθυντής, ε, αναπληρωτής της DG DEFCO, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής και θα μας μιλήσει για τον, τον ρόλο της Αφρικανικής Διασποράς στην Ευρώπη, για την ανάπτυξη της Αφρικής, αλλά και θα μας μιλήσει και για τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Κατόπιν θα δώσω το λόγο απευθείας στους προσκεκλημένους, ξεκινώντας από την κυρία Μάνκε. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όλοι μαζί οι ομιλητές έχετε 30 λεπτά συνολικά. Η κυρία Μάνκε λοιπόν από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, άρα το πολύ 10 λεπτά σας παρακαλώ, γιατί όπως σας είπα συνολικά θα ε, διαρκέσουν οι ε, ομιλίες σας 30 ε, λεπτά. Καλησπέρα, Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που... Χαίρομαι που συμμετέχω σε ένα πάνελ διακεκριμένων ομιλητών που θα παρουσιάσουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Η παρουσία PowerPoint ε, που είχα ετοιμάσει ακριβώς για να σας δώσω τις τάσεις ε, και άλλα στοιχεία δυστυχώς δεν μπορεί να προβληθεί, λυπούμε. Ελπίζω και αυτά που σας είπα να είναι εξίσου ενδιαφέροντα με αυτά που θα βλέπετε στις διαφάνειες. Για να έχετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα σε ό,τι αφορά την Αφρικανική Διασπορά επιτόπου, εν συντομία μου ζητήθηκε να μιλήσω για ένα θέμα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα. Να κάνω μια εισαγωγή και μετά να μπω σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Η διασπορά είναι εταίρος ανάπτυξης ε, για την ε, υλοποίηση του Παγκόσμιου Συμφώνου Μετανάστευσης αλλά μας βάζει και σε προοπτική γενικά για την Αφρική. Να ξεκινήσω με κάποια βασικά μηνύματα. Το πρώτο, νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε και γνωρίζουμε το ιστορικό πλαίσιο. Η ιστορική στιγμή είναι ακριβώς η έγκριση, ελπίζουμε, του Παγκόσμιου Συμφώνου για την νομότυπη μετανάστευση. Το έχω βάλει και στον τίτλο της παρουσίασής μου τα άτομα, οι μετανάστες, η κοινότητα των πολιτών είναι οι εταίροι, πραγματικοί εταίροι της ανάπτυξης. Εμείς εργαζόμαστε για δεκαετίες ως οργάνωση στον τομέα αυτό. Στηρίζουμε κυρίως τις κυβερνήσεις, εταίρους διαφόρων μερών της κοινωνίας γιατί θεωρούμε ότι για να υπάρξει μια σωστή αντίληψη κινητικότητας και μετανάστευσης δεν πρέπει να τονίζουμε το σκέλος ε, της ασφάλειας, αλλά πρέπει να συζητήσουμε και για άλλα θέματα της μετανάστευσης και της κινητικότητας, ότι δηλαδή πραγματικά διευκολύνουν και προωθούν ε, την ανάπτυξη. Αυτό είναι το μήνυμα που ε, στέλνει η δική μας οργάνωση. Δυστυχώς όμως δεν ακούγεται επαρκώς το ίδιο κίνημα, με μήνυμα στην κοινωνία. Πρέπει να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτό το μήνυμα. Όταν μιλάμε για γενικές ιδέες και έννοιες, δεν μπαίνουμε στην ουσία. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να μιλήσει κανείς θετικά για την κινητικότητα. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να εξηγήσει κανείς ε, τη θετική πλευρά της μετανάστευσης. Διότι πολύ συχνά κινητικότητα μετανάστευση συνδέονται με το έργο που κάνουμε επί τόπου, Υπουργείο Εσωτερικών και πιο πολύ με το ρυθμιστικό σκέλος. Η κινητικότητα όμως είχε γκάρσια φύση. Δηλαδή, εντάσσεται στις οικονομικές δραστηριότητες, ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί, αλλά έχει να κάνει και με κοινωνικά ζητήματα, έχει να κάνει με περιβαλλοντικά ζητήματα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, όλες τις πτυχές και κάθε μέρος της δίκης της κυβέρνησης ε, και οι βουλευτές πρέπει να συμμετέχουν. Είναι καλό που το συζητάμε εδώ ε, στον οίκο των Ευρωβουλευτών. Διότι για μας το Κοινοβούλιο είναι ένας εταίρος. Οι βουλευτές πρέπει να είναι στο πλευρό μας αν θέλουμε να αναπτύξουμε αποτελεσματικές μεθόδους για την διαχείριση της κινητικότητας και το Παγκόσμιο Σύμφωνο ακριβώς για αυτό το σκοπό θέλουμε να ε, ιδρυθεί. Λοιπόν, θα, θα μιλήσουμε για τις διασπορές εν γέννη. Έχω φέρει κάποια στοιχεία. Είναι ένα θέμα που δύσκολα μπορεί κανείς να το αναπτύξει. Τι τάσεις υπάρχουν λόγω των στοιχείων που έχουν στη διαδεσία μας για μετανάστευση. Καταλαβαίνετε το λόγο, αλλά θα σας εξηγήσω και από πλευρά μου. Προσπαθούμε να καταγράψουμε αυτούς οι οποίοι μετακομίζουν ε, ή διαμένουν κάπου ε, αλλού, σε κάποια άλλη χώρα. Αλλά η διασπορά είναι ένας ε, όρος πολύπλοκος. Ανάλογα με την χώρα και την κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιείται άλλη ένωση, να υπάρχουν άλλη, συνειρ... άλλη ορολογία, άλλη έννοια, να υπάρχουν άλλοι συνειρμοί σε ό,τι αφορά την έννοια διασπορά. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να καταλήξει κανεί σε κάποιε παγκοσμίε Θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε για αριθμού τη διασπορά Συνήθως αναφερόμαστε σε εκτιμήσεις ε, για τους διεθνούς μετανάστες. 258 εκατομμύρια διεθνείς μετανάστες, αυτός είναι ο αριθμός που έχει υπολογιστεί. Αυτό το χρησιμοποιούν ε, το νούμερο διάφορες οργανώσεις όπως είναι ο ΣΑ, για παράδειγμα, όταν θέλουν να λύσουν ε, τάσεις και να δώσουν κάποια χαρακτηριστικά. Ε, στη, στους μετανάστες, τι επίπεδο δεξιοτήτων, τη γνώση, σε ποια είναι η χώρα τα κτλ. Αυτό που λείπει όμως είναι το εξής. Η διασπορά περιλαμβάνει και την έννοια της, ε, των μεταναστών δεύτερης γενιάς, όπως τους λέμε. Κάποιες χώρες, σε κάποιες κοινωνίες υπάρχει έννοια της ε, ηθικής ενότητας, η διασύνδεσης και εμείς στην οργάνωσή μας την διασπορά την ορίζουμε ως τις οργανώσεις εκείνες που έχουν ε, ε, ισχυρού δεσμούς με τη χώρα καταγωγής τους, χώρα προέλευσης. Συνολικά λοιπόν πολύ δύσκολο να κάνει κανείς λόγο για τάσεις, πόσο μάλλον να τις ανοιχνεύσει. Προσπαθούμε πάντως. Στις διαφάνειές μου θα μπορέσω ίσως να σας στείλω την παρουσίαση ηλεκτρονικά. Είχα κάποια γραφήματα για να δούμε ποιες είναι οι κύριες χώρες προέλευση μεταναστών στην Αφρικανική Ήπειρο και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι περισσότεροι μετανάστες είναι Αίγυπτο, Μαρόκο, Σομαλία, Σουδάν, Αλγερία και... Εδώ μιλάμε για ένα εκατομμύριο τουλάχιστον μετανάστες που φεύγουν τις χώρες αυτές και πάνε στο εξωτερικό. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την Αφρική και το, τη μετανάστευση, πολλή κινητικότητα ε, υπάρχει και εντός της Υπήρου, προσωρινή κινητικότητα. Αλλά αν δείτε και τους αριθμούς μεταναστών, το 80% περίπου των μεταναστών γεννιούνται σε μια χώρα και πηγαίνουν σε μια άλλη αφρικανική χώρα. Αν υπολογίσουμε τα στοιχεία του ΟΕΕ για τους μετανάστες, έχουμε 36 εκατομμύρια και πάνω, οι οποίοι πηγαίνουν σε κάποια χώρα της Αλοδαπή. Στο γράφημα υπήρχαν και κάποιες τάσεις ε, το της τελευταίας μας έκθεσης, ε, της έκθεσης της περσινής χρονιάς, βλέπαμε την κινητικότητα εκεί και προς την Ευρώπη, γιατί θέλαμε να δούμε ποιες είναι οι κινήσεις προς την Ευρώπη και εκεί καταγράφηκε αύξηση, αλλά και άλλες Ήπειροι και άλλες ε, χώρες καταγράφουν αντίστοιχε τάσει. Υπάρχουν προκλήσει για την περιγραφή του φαινομένου. Εμεί εργαζόμαστε σκληρά για να στηρίξουμε το κυβερνητικό έργο και το έργο των άλλων εταίρων. Ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιες είναι οι λύσεις, πώς ε, ε, εστιάζουμε στις πρακτικές για να δούμε και τι αντίκτυπο έχουμε επί τόπου. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα και εταιρικέ σχέσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου. Για παράδειγμα, αν δούμε τα περσινά νούμερα, κατά τουλάχιστον γραφεία έχουμε ε, και εργαζόμαστε για τα θέματα της διασποράς, στηρίζουμε την ανάπτυξη πολιτικών ε, από την κυβέρνηση ή σχεδιάζουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Πώς στηρίξαμε τις μελέτες, μάλλον τα τελευταία πέντε χρόνια κάναμε κάποιες μελέτες, 150 τον αριθμό. Diaspora Mapping, ε, χαρτογράφηση διασποράς, έτσι είναι ο τίτλος αυτών των μελετών. Υπάρχουν διάφορα έργα και πρωτοβουλίες. Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της μεθοδολογίας ε, για τη διεξαγωγή των χαρτογραφήσεων και μελετών αυτών. Και εμείς και άλλες οργανώσεις κάνουμε τέτοιου μελέτες. Το 2013 σε υπογικό επίπεδο συζητήθηκε το θέμα της ε, διασποράς ε, γιατί έχει προσλάβει μεγάλη σημασία στο γενικότερο θεματολόγιο και μαζί με ομολόγους από το Συμβούλιο της Ευρώπης οργανώσαμε ε, κάποιες ε, εκδηλώσεις στη Γενέβη για την ε, συμμετοχή της διασποράς και το συμπέρασμα ήταν ότι η νόμη, η ρύθμιση πρέπει να ληφθεί υπόψη για να έχουμε ένα περιβάλλον που θα διευκολύνει τη συμμετοχή της διασποράς. Βέβαια, το πρόβλημα δεν είναι συνήθως ο νόμος, όχι ότι δεν είναι σημαντικό, βέβαια, αλλά σημαντικό είναι να στηριχθούν οι πρωτοβουλίες και να υπάρξει ένα έφορο, ένα γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλειών. Κάποια από τα προγράμματα που είναι σημαντικά για εμάς, ένα από αυτά είναι το Migration for Development in Africa. Σε συνεργασία με διάφορες κυβερνήσεις όπως το Βέλγιο, η Ιταλία αναπτύσσουμε τέτοια προγράμματα και η Φιλανδία συμμετέχει προσφάτως για τους επαγγελματίες που παραδείγματος ε, επανέρχονται στη χώρα του στην Σομαλία, στην προκειμένη περίπτωση και εργάζονται στον τομέα της υγείας. Ε, θέλουμε επίσης να αναφέρουμε και την ε, Ολλανδική κυβέρνηση. Υπάρχουν εκπρόσωποι της Διασποράς ε, και προωθούν κάποιες πρωτοβουλίες επιτόπου. Τρεις είναι Τρία παραδείγματα θα σας δώσω. Πώ um, Πώς μπορεί η Διασπορά να μας βοηθήσει εργαστούμε στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, του εμπορίου, των επενδύσεων. Έχουμε μια περίπτωση, δημιουργήθηκαν κάποια δίκτυα ε, πληροφορικά συστήματα στον τομέα της υγείας ή μια άλλη πρωτοβουλία είναι υποστήριξη ειρηνευτικών προσπαθειών από τη Διασπορά. Ένα γραφείο που έχει έδρα στην Αμερική βοηθά προγράμματα για να υπάρχει ένα είδος ανθεκτικότητας για καταφυγίων, καταβλισμών για χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Στη Σομάλιλαντα, αλία, εκπαίδευση. Εκεί η διασπόρα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά επιτόπου. Έχει μεγάλη σημασία να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια. Είπα ότι συνήθως δίνουμε δεσπόσα σημασία στην ασφάλεια και τη ρύθμιση. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε από κοινού οι διάφορες οργανώσεις. Και εμείς σε λίγες εβδομάδες θα δρομολογήσουμε μία πύλη για τη διασπορά. Στόχος είναι εκεί να συγκεντρώσουμε την εμπειρία όλων των σχετικών οργανώσεων, εκμεταλλευόμενοι και το δίκτυο που έχουμε επί Αυτή η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή είναι υποκατασκευή και παίρνουμε feedback. Υπάρχει ένα συμβουλευτικό ε, νομοθετικό συμβούλιο, εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού κόσμου. Η Diaspora είναι στο Google ο σύνδεσμος και εκεί μπορείτε να δείτε 8 Οκτωβρίου Διεθνής Διάλογος για τη Μετανάστευση. Κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είπα ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε, να εργαστούμε μαζί. Διαρκής είναι και η συγκέντρωση δεδομένων, οι κοινέ προσεγγίσει, αλλά και οι συμπράξει εταιρικέ σχέσει στον τομέα του Παγκοσμίου Συμφώνου. Θα γίνουν πολλά, θα υπάρχουν πολλέ δυνατότητε και ευκαιρίε. για δημιουργία υποδομών, δυνατοτήτων, θα υπάρχει σχετικό μηχανισμό. θα έχουμε μια πλατφόρμα ανταλλαγή πληροφόρων και γνώσεων. Και εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ. Merci euh. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάνκε. Σας ευχαριστούμε γιατί θα σας έκανα και νόημα ότι είχε ολοκληρωθεί ο χρόνο αγορευσή σα. Είχατε υπερβεί λίγο τα 10 λεπτά, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέγατε. Πρέπει να σα πω ότι αναφερθήκατε σε πολλά ενδιαφέροντα σημεία και όσοι μα ακούνε σίγουρα θα μπορούν στη συνέχεια να θέσουν τυχόν ερωτήσει και πρέπει να σα πω ότι η συνεδρίασή μα μεταδίδεται και μέσω του διαδικτύου. Υπάρχει λοιπόν και ένα κοινό το οποίο μα ακολουθεί μέσω του διαδικτύου πέρα από την αίθουσα αυτή δηλαδή. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για όλα τα σημεία που θίξατε και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ντιόπα ο οποίο είναι σύμβουλο, στην εταιρεία συμβούλων Schumann Associates και ασχολείστε ιδιαίτερα με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ιδιωτικέ επενδύσεις, τη μετανάστευση και τη διασπορά. Σας δίνω για πέντε περίπου λεπτά το λόγο, αλλά σε κάθε περίπτωση, μην ανησυχείτε, θα έχετε την ευκαιρία να δευτερολογήσετε, θα απαντήσετε σε ερωτήσει. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας, για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συμμετέχω στην πολύ σημαντική αυτή ακρόαση που θεωρώ ότι λαμβάνει χώρα την κατάλληλη στιγμή. Καθότι θα μιλήσουμε για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Αφρικανική Διασπορά και πώς μπορεί να συμβάλλει στην απτεξική πολιτική που προωθεί στην Αφρικανική Ήπειρο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και 10 χρόνια περίπου στα πλαίσια των Schumann Associates, τη εταιρεία αυτή συμβούλων, εργάζομαι για τα ζητήματα αυτά, αλλά δραστηριοποιούμε επίση και στην ε, Σενεγάλη μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλειών που έχουν να κάνουν με προγράμματα πρόσβασης ε, στην υγεία, στον οικογενειακό προγραμματισμό και το καθεξής. Θα αναφερθώ στα ζητήματα αυτά στο τέλος παρουσίασής μου. Πώ μπορεί να εμπλακεί περισσότερο η Αφρικανική Διασπορά στην Ευρώπη στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασία. Η διασπορά αυτή είναι μια δύναμη δημογραφική αλλά και οικονομική θα ήθελα να ξεκινήσω με την οικονομική αυτή πτυχή, δίνοντά σα κάποια αριθμητικά δεδομένα. Ένα μάλιστα αριθμητικό δεδομένο που θα μα επιτρέψει να καταλάβουμε πραγματικά πόσο σημαντική είναι αυτή η οικονομική πτυχή. 65 δισεκατομμύρια δολάρια. 65 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το ποσό των εμβασμάτων που γίνονται από την Ευρώπη προ την Αφρική, από την Αφρικανική Διασπορά προ την Αφρικανική Ήπειρο και αυτό μόνο και μόνο για το 2017 και ουσιαστικά είναι ένα ποσό το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια που αποτιμάται περίπου στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ε, πάνω από το 50, ένα 50% του ποσού αυτού είναι κυρίως ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία πηγαίνουν προς την Αφρική και τα περισσότερα βέβαια από τα κονδύλια αυτά έχουν να κάνουν με καθημερινές δαπάνες υγείας, ε, Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα, δαπάνες στέγαση, και Όλα αυτά τα σημεία θα τα καλύψω αργότερα. Επειδή υπάρχει και η δημογραφική πτυχή. Η Αφρικανική Ένωση αναφέρεται στην Αφρικανική Διασπορά ως την έκτη περιφέρεια της Αφρικανικής Υπήρου και η Αφρικανική αυτή διασπορά κατανέμεται με τον ακόλουθο τρόπο. Περίπου 112 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται στη Λατινική Αμερική, 39 εκατομμύρια στη Βόρεια Αμερική, 13 εκατομμύρια στην περιοχή της Καραϊβικής και όσον αφορά την Ευρώπη έχουμε περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια άτομα, πολύ λιγότεροι δηλαδή είναι παρόντες στην Ευρώπη από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ποιε είναι οι βασικέ χώρε υποδοχή, προφανώ η Γαλλία με πάνω από το 50%, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία και οι κάτω χώρε. Μολονότι ε, η σημασία η οικονομική και δημογραφική της Αφρικανικής Διασποράς είναι πολύ σημαντική και διόλου αμεληταία. Η παρουσία της και η βαρύτητα της διασποράς όσον αφορά την ανάπτυξη, όσον αφορά τις πολιτικές μετανάστευσης, όσον αφορά την επένδυση, δεν προβάλλεται τόσο πολύ. Πώς μπορούμε λοιπόν στο υφιστάμενο αυτό πλαίσιο, όπου βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αναδιαρθρώσει τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής, μέσω της οικονομίας. Πριν από δύο περίπου εβδομάδες ο πρόεδρος Γιούνκερ μιλώντας για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μίλησε όλο και περισσότερο για τις επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν, για το εμπόριο, αλλά, και για την ε, κατάρτιση των ε, Αφρικανών, καθώς επίσης και την ε, δημιουργία πολλών θέσεων απασχόλησης μέχρι το 2020. Και μην ξεχνάμε ότι έχουν επίσης και όλα αυτά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία όλο και περισσότερο συνδυάζουν δημόσιες και ιδιωτικέ επενδύσεις. Είχα αναφερθεί στα ζητήματα αυτά και σε ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, όπου έλεγα ότι πραγματικά θα έπρεπε ο ιδιωτικό τομέα να προωθηθεί ακόμα περισσότερο στο πλαίσιο τη επενδυτική αυτή πολιτική. Πιστεύω λοιπόν ότι στον ιδιωτικό αυτό τομέα μπορεί πραγματικά να δραματίσει από οικονομική πλευρά ένα πολύ σημαντικό ρόλο η Αφρικανική Διασπορά, η οποία μπορεί να προωθήσει σαφώ επενδύσει αυτέ, αλλά μπορεί να συμβάλλει στο να έχουν μεγαλύτερη παρουσία οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Αφρικανική Ήπειρο, να συμμετέχουν και αυτές όλο και περισσότερο σε επενδυτικά προγράμματα. Πώς μπορούν λοιπόν να συμμετέχει όλο και περισσότερο σε τέτοιες πρωτοβουλίες η Αφρικανική Διασπορά. Ξέρετε ότι γίνονται ήδη κάποιες αναφορές όσον αφορά τα εθνικά ετήσια προγράμματα, τα επενδυτικά, τα πολιετή προγράμματα, τα επενδυτικά τα οποία λαμβάνουν χώρα. Θα μπορούσαμε να βρεθούμε επίση στα διεθνή φόρα τα οποία προωθούν οικονομικέ επενδύσει προ την Αφρικανική Ήπειρο. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε επίση και για τα προγράμματα κατάρτιση, για το mentoring, την καθοδήγηση. Θεωρώ όμω ότι το πιο σημαντικό είναι να δούμε τι υφίσταται αυτή τη στιγμή επί τόπου, τι λειτουργεί σωστά και πώ μπορούμε ουσιαστικά να πολλαπλασιάσουμε τη θετική αυτή επίδραση των υφιστάμενων προγραμμάτων και πρωτοβουλειών. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω πολύ γρήγορα, κυρία Πρόεδρε, αναφερόμενο στην μη κυβερνητική οργάνωση για την οποία εργάζομαι, την μη κυβερνητική οργάνωση ΡΑΕΣ, στην οποία εργάζομαι από το 2014. Εδώ χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως στην τηλεόραση. Αρχίσαμε με το ραδιόφωνο, αλλά τώρα επεκτεθήκαμε και στην τηλεόραση και ουσιαστικά θα ήθελα να αναφερθώ σε μία τηλεοπτική σειρά η οποία ονομάζεται Σελαβή, έτσι είναι η ζωή, και η οποία προβάλλεται αυτή τη στιγμή σε 26 χώρες με πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους που την παρακολουθούν. Στα πλαίσια της σειρά αυτή δίνουμε όλο και περισσότερο το λόγο στους νέους και στα 36 επεισόδια του πρώτου και του δεύτερου κύκλου καλύπτουμε διάφορα ζητήματα τα οποία πολλές φορές είναι ακόμα ταμπού χωρίς εμεί να υποδεικνύουμε τι πρέπει να κάνει ο καθένας αλλά δίνοντας την ευκαιρία στους νέους αυτούς να αρχίσουν να μιλάνε ελεύθερα για όλα αυτά τα ζητήματα. Και έχουμε δημιουργήσει επίση και εταιρικέ σχέσει μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και οι νέοι από την Αφρική αλλά και οι Αφρικανοί οι οποίοι συμμετέχουν στην Αφρικανική Διασπορά και βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχουν στο να δημιουργηθεί τηλεοπτικό περιεχόμενο, αν θέλετε, προκειμένου να καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον τοπικό πληθυσμό στην Αφρική, κυρίω του νέου στα σχολεία. Χρησιμοποιούμε, όπω βλέπετε, όλο και περισσότερο τι νέε τεχνολογίε, τα μέσα κοινωνική δικτύωση, το Facebook και όλα τα άλλα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν όλο και περισσότερο οι νέοι και συνεργαζόμαστε και για μία άλλη τηλεοπτική σειρά, η οποία θα φέρει τον τίτλο «Bruit de tambour», ο ήχος των τυμπάνων. Η σειρά αυτή θα αναφέρεται όλο και περισσότερο σε πολιτικά ζητήματα, στη συμμετοχή στα κοινά, στην ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Ξέρετε ότι το ζήτημα των εκλογών, οι προεκλογικέ εκστρατείε είναι πολλέ φορέ ζήτημα ιδιαίτερα ευαίσθητο στην Αφρική και θέλουμε ακριβώ να ευιστοποιήσουμε περισσότερο του νέου για μία συμμετοχή σε ένα ευνοϊκό θετικό κλίμα, στη συμμετοχή ε, σε έναν τέτοιο διάλογο μεταξύ των διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα το οποίο τελικά θα συμβάλλει στο να αλλάξουν οι νοοτροπίε. Πρέπει να σας πω ότι ο ρόλος της διασποράς για μένα θα είναι πραγματικά να γίνει η φωνή τη Ευρώπη όσον αφορά την Αφρική, προωθώντα την Αφρική δηλαδή τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώ για το λόγο αυτό τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστούν περισσότερο με την Αφρικανική Διασπορά στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Διόπ. Τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε εδώ είναι πολύ ενδιαφέροντα, κυρίως όμως τα θέματα που θίξατε, αλλά και τα ε, προγράμματα. Μιλώντας για την διασπορά ως την έκτη περιφέρεια της Αφρικανικής Υπήρου και τώρα δίνω τώρα το λόγο σε μια άλλη κυρία, ε, στην κυρία Μαρή Σοντάλ που είναι διευθύντρια του ADNE και πρόεδρος του, πρόεδρο του Δικτύου Αφρικανικής Διασποράς ε, στην Ευρώπη. Μαρίσον Τάλ, αν δεν κάνω λάθος, θα μας εξηγήσει τα θέματα αυτά. Ε, θα σας ε, ξανασυναντηθούμε εδώ στο Κοινοβούλιο στις 5 Οκτωβρίου, που οπότε θα ξεκινήσει η Εβδομάδα Παγκόσμιας Διασποράς. Η Μαρίσον Τάλ θα μας αναπτύξει αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ. Θα ήθελα ξεκινώντας να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου τη, στην κυρία Κέγκε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία οργάνωσε μια συνεδρίαση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Θεωρώ ότι αυτή η ακρόαση ε, επιβεβαιώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί και τη φωνή όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Οι πολίτες μας, οι χώρες μας δυναμώνουν αν ε, ε, υιοθετήσουμε την πολυμορφία και ακούγονται όλες οι φωνές, ακόμα και η φωνή της διασποράς. Ε, για τη διασπορά μίλησαν οι προλαλήσαντες. παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση της φτώχειας, στην ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη των χωρών, χωρίς βεβαίως να ξεχνάμε τη συνεισφορά της χώρες υποδοχής. Ο φίλος μου αναφέρθηκε στο ότι τα χρήματα που στέλνει διασφορά είναι περισσότερα από τα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά κονδύλια. Ε, ε βεβαίως ε, αυτά επέτρεψαν την πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση των παιδιών, όπως επίσης και την ανάπτυξη ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή βιομηχανιών αυτά που είπε ο κύριος Διόπ δείχνουν ότι παρά τη σημαντική αυτή συνεισφορά η διασπορά μένει στο περιθώριο ως παράγοντας ανάπτυξης τόσο στις συζητήσεις όσο και στις πρωτοβουλίες. Αυτή η δυσάρεστη διαπίστωση μας ε, προκάλεσε την ιδέα δημιουργίας ενός δικτύου αφρικανικής διασποράς στην Ευρώπη το 2015. Το 2015 ήταν σημαντική χρονιά για την ανάπτυξη, η συνεργασία για την ανάπτυξη, γιατί ήταν ε, το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης, αλλά και το έτος όπου υιοθετήθηκε το αναπτυξιακό θεματολόγιο του για το 2030. Ξεκίνησαμε λοιπόν ε, τις εκστρατείες για την βιώσιμη ανάπτυξη και αποφασίσαμε να θεωρηθεί ο πολιτισμός εργαλείο ανάπτυξης. Όπως γνωρίζετε, από μόνη της η ανάπτυξη είναι μια έκφραση. Η κατανόηση της γραφής και του κοινωνικού πλαισίου ε, των ε, χωρών της ανάπτυξης είναι σημαντικές για την ε, κατανόηση των ε, αναγκών και του πλαισίου σε τοπικό επίπεδο. Και βεβαίως η διασπορά ανήκει και στους δύο κόσμους. Γνωρίζει και το πλαίσιο της χώρας προέλευσης αλλά και το, την τεχνογνωσία της χώρας υποδοχής, πράγμα που μας επιτρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί ε, στον τομέα της πρόθεσης ανάπτυξης. Ε, προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά διευκολύνοντας τη συμμετοχή της διασποράς στις αναπτυξιακές προσπάθειες ε, με τη δημιουργία μέσων για την εκμετάλλευση αυτού του ανεκμετάλλευτου δυναμικού της διασποράς ε, στην προσπάθεια πλαισίωσης των νέων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και συνεργασίας στις χώρες προέλευσης. Σήμερα ε, εκπροσωπώ μια, ε, μια οργάνωση που περιλαμβάνει πάνω από 40 ε, οργανώσεις στην Ευρώπη. Το δίκτυο αυτό επέτρεψε την δημιουργία στρατηγικού διαλόγου και εταιρική σχέσης ανάμεσα στις οργανώσεις και των ε, θεσμικών οργάνων. Ανήκουμε στο Policy Forum for Development που ε, εκπροσωπείται η κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης αλλά και όλες οι ομοσπονδίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη. Είναι ένα σημαντικό βήμα και θα ήθελα γι' αυτό να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία επέμεινε να εμπλακεί η διασπορά εκεί σε αυτή τη διαβούλευση. Επίσης, ε, συμμετείχε στη διάσκεψη κορφής της Βαλέτας για την μετανάστευση με συστάσεις για τη διασπορά και παρακολουθώντας την εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης πρέπει να πω ότι σήμερα παρά τις καλές προθέσεις της διάσκεψης κορφής της Βαλέτας ε, εξακολουθούμε να, ε, να, να να παραμένουμε ως διασπορά στο περιθώριο και αν δεν μας χρησιμοποιούν στην, ως δυνατότητα εξέβρεσης ε, λύσεων ε, στον τομέα αυτό. Δηλαδή τα λόγια δεν έγιναν πράξη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποιες πρωτοβουλίες που ξεκινήσαμε και που υλοποιούμε στο πλαίσιο του δικτύου μας στην Ευρώπη για να διευκολύνουμε τη συνεργασία με τις χώρες υποδοχής και τα θεσμικά τους όργανα. Δουλεύουμε για τη δημιουργία ε, μια βάση δεδομένων, την African Diaspora Skills Database, η οποία ενημερώνει για τα ενδιαφέροντα της διασποράς όσον αφορά τις επενδύσεις αλλά και την απασχόληση ώστε να μπορέσει να πλαισιωθεί το κίνημα επιστροφής και της ε, ανταλλαγής γνώσεων, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας με τις χώρες της υποδοχής. Τέλος, όπως είπε και η κυρία Κέγγελ, ε, εδώ από το 2015 ε, έχουμε ε, γιορτάσει την Ευρωπαϊκή ε, Εβδομάδα Διασποράς. Ε, γίνονται εκδηλώσεις και στις χώρες υποδοχής αλλά και στις χώρες προέλευσης, αλλά καταδικάζουμε και τον, τις διακρίσεις κατά των μεταναστών, γιατί η κατανόηση της διασποράς είναι σημαντική, γιατί πολύ συχνά γίνεται σύγχυση μεταξύ οικονομικών μεταναστών και ε, ε, μεταναστών ε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε ποιον απευθυνόμαστε. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις 5 Οκτωβρίου θα ξαναέρθουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, το πρόεδρο του Κοινοβουλίου που επέκτηνε την επίσημη ε, πρόσκληση ε, ή μας έθεσε υπό την αιγίδα ούτω ώστε την, να επιτύχουμε τους σημαντικούς στόχους. Θα κλείσω ε, αναφερόμενοι σε τρεις-τέσσερις συστάσεις, όπως το στόχος του να εμπλακεί η διασπορά στην υλοποίηση των στόχων της ανάπτυξης. Ε, έχουμε πέντε συστάσεις που αφορούν τα μέσα, που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε αυτή την ε, εμπλοκή. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα που θα γίνονται ανταλλαγές ε, με τη διασπορά, με τρόπο διαρθρωμένο. Επίσης, ε, να εμπλέκεται η διασπορά τις ε, συζητήσεις που γίνονται ε, εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η ακρόαση είναι σημαντική για το σκοπό αυτό, να επιμένουμε στην δυσκολία πρόσβασης στους πόρους και στα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται για τη διασπορά παίζει σημαντικό ρόλο, ή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο η διασπορά, αλλά αν δούμε το χάρτη ε, πού βρίσκονται οι οργανώσεις της διασποράς. Πρέπει να κάνουμε τα λόγια πράξη. We need to walk the talk, όπως λέμε στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci beaucoup. Σας ευχαριστούμε. Μαρή σας ευχαριστούμε για όλες αυτές τις πληροφορίες. Θα επανέλθουμε αργότερα. Και τώρα θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον τελευταίο μας ομιλητή, τον Hans Στάουσμπολ από τη ΓΔ Ντεύκο. Σειρά σας να πάρετε το λόγο για να μας εξηγήσετε τι πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά αυτές τις δράσεις που έχουν επίκεντρο την Αφρικανική Διασπορά για μια πιο αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία στην Αφρική. Θα μας παρουσιάσει την κυρία Στάσμπο λοιπόν τις βασικές θέσεις της ε, Ένωσης, της Κομισιόν για αυτές τις πρωτοβουλίες, για αυτά τα προγράμματα που είναι πολύ άριθμα και είμαι βέβαια ότι έχετε επιλέξει τα πιο σημαντικά για το κρατήριό μας. Ελπίζω να μην παραλείψετε να μιλήσετε για μία από τι πιο πρόσφατε δράσει που είναι η στήριξη ενό μέσου διευκόλυνση ε, στο πλαίσιο της ετή, του ετήσιου προγράμματος, ε, το θεματικό πρόγραμμα για τα παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Η οικονομική συνεισφορά αναλαμβάνεται από την Ένωση στο πλαίσιο του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας. Έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τρία λεπτά βλέπω ότι μου έχουν μείνει περίπου, αλλά τέλος πάντων ε, οι προλαλήσαντες έχουν αναφέρει τα βασικά ζητήματα και ήδη ακούστηκαν και κάποιες συστάσεις. Για να πλαισιώσω το θέμα, θέλουμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να τους συμπεριλάβουμε ε, στις προσπάθειες να γνωρίσουμε τι διασύνδεσει μετανάστευση και ανάπτυξη. Μπορεί να έχει ένα θετικό ρόλο στην ανάπτυξη μετανάστευση. Για μα, βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο και στην αναπτυξιακή μα πολιτική το θέμα τη μετανάστευση μα απασχολεί εδώ και χρόνια και σε ό,τι αφορά τι προκλήσει αλλά και σε ό,τι αφορά τι ευκαιρίε που προσφέρει. Και σε αυτό το πλαίσιο, η διασπορά είναι ένα μέρο τη προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως ε, είπαν οι προλαλήσαντες, αναφέρεται και στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ε, εφτακτή ασφαλή ε, νομότυπη μετανάστευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος για τη συμμετοχή των διασπορών στον πληθυντικό στους της βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχος είναι το κόστος να υποστημίωσε κατά 3% και θέλουμε να κλείσουμε επίσης ε, κάποιους ε, ακριβούς διαδρόμους. Θέλουμε το στόχο αυτό να τον πετύχουμε και είναι μια δέσμευση που στο κοινό σχέδιο δράσης που είπε η Στάφος Εξεγονίμων ε, προηγουμένως. Ήδη έχουμε να αναλάβει περαιτέρω δεσμεύσεις. Μέχρι το 2030 θέλουμε να έχουμε εντοπίσει χώρες εταίρες που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας σε θέματα που αφορούν το τη μείωση του κόστου βιώσιμη ανάπτυξη που έχουμε εντοπίσει στου διαδρόμου. Πρέπει να συνεργαστούμε και με τον ιδιωτικό τομέα και με άλλου, όπω και με τη διασπορά. Εδώ και χρόνια με τη διασπορά προωθούμε τον περιφερειακό διάλογο σε διάφορους τομείς. Από το 2006, μαζί με τους Αφρικανούς εταίρους, βλέπουμε ποιος είναι ο ρόλος της διασποράς σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τη μετανάστευση. Σημαντική ήταν η προσπάθειά μας ε, για την κατάρτιση του σχεδίου δράσης του Μαρακές το Μάιο του 2008 και εκεί φαίνεται πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος για, την, για τις χώρες προέλευσης, ε, διέλευσης και προορισμού. Το ρόλο παίζει η Διασπορά. Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία με τη Διασπορά. Όπως είπε και η Πρόεδρος, από το 2016 στηρίζουμε και κάποια προγράμματα στον τομέα αυτό. Όλες τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Θα σας δώσω κάποια. Το Μετάφρικα, το African Invest, για την ε, Βορειοδυτική Αφρική, το MedWest Africa και στο πλαίσιο του διαλόγου για τη μετανάστευση και την κινητικότητα μεταξύ Ένωσης και Αφρικής Έχουμε στηρίξει δρομολόγηση με πρωτοβουλίων το 2015 και εφαρμόζουμε σχετικά κάποιες δράσεις. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι τον Νοέμβριο πέρυσι έγινε η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής και είπαμε ότι η Διασπορά είναι βασικός εταίρος στην όλη διαδικασία. Έχουμε το καταπίστευμα για την Αφρική στηρίζουν στο πλαίσιο αυτού πολλές πρωτοβουλίες στη Δυτική Αφρική, σε χώρες όπως Νιγηρία, Μαυριτανία και Σενεγά. Να μην πω σε λεπτομέρειες τώρα. Βέβαια, στηρίζουμε τις χώρες εταίρους και τις περιοχές οργανώσεις ε, για την καλύτερη διαχείριση της κινητικότητας και τη μετανάστευση συνεργασία μέσω ομολόγων. Παρέχουν προσαρμοσμένη εξατομικευμένη βοήθεια κατόπιν ετήματος. Έχουμε το πρόγραμμα το ειδικό για την ε, μετανάστευση και παρέχουμε εμπειρία και τεχνογνωσία. Στο Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Πρόγραμμα και σημείωσα αυτό που είπε ο συνάδελφος εκ δεξιών, ένα από τα πρώτα προϊόντα, αν θέλετε, που εντοπίσαμε στη νέο μέσο ε, εγγύησης, έχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Inclusive 5, ένα πρόγραμμα εγγύσεων για κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου με στόχο τη διασπορά για να μπορέσουν ε, οι Αφρικανοί αλλά και οι χώρες της γειτονίας ε, να παίρνουν ε, χρηματοδότηση πιο εύκολα. Θέλουμε να υπάρξει προσέλκυση επενδύσεων από τη διασπορά, επενδύσεις σε επιχειρήσεις που έχουν γίνει από ντόπιου και τις οικογένειές τους και θέλουμε να βοηθήσουν και οι διάφοροι φορείς και να δώσουν ευκαιρίες. Αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η διασπορά και θέλουμε να βρούμε νέου τρόπου για να προωθήσουμε στρατηγικό διάλογο, εταιρικέ σχέσει. Οπότε το Μάρτιο φέτο οργανώσαμε ε, μια ομάδα ε, για ε, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στο πλαίσιο τη επιτεύξης των στόχων στρατηγικής ανάπτυξη με συμμετοχή τη Διασπορά. Προτείνουμε επίση ένα νέο μέσο διευκόλυνση, το οποίο μάλλον θα συζητηθεί αύριο στην Επιτροπή DCI, με το Συμβούλιο. Είναι ένα νέο πρόγραμμα που λέγεται Support for Global Youth Diaspora Facility. 5 εκατομμύρια ευρώ είναι ε, το κονδύλιο του προπολογισμού για αυτό το πρόγραμμα θέλουμε οι οργανώσεις της Διασποράς των χωρών καταγωγής να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά. Τέσσερις συνιστώσεις, παγκόσμια χαρτογράφηση για την συμμετοχή της διασποράς, δημιουργία υποδομών και τεχνική βοήθεια για κυβερνήσει και των πολιτών και οργανώσεις της διασποράς, πλατφόρμα για ένα διαθρωμένο διάλογο και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα δίκτυο εμπειρογνωμών από τη Διασπορά που θα παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία. Αύριο στην Επιτροπή DCI ελπίζουμε να το εγκρίνουν τα κράτη-μέλη και έτσι θα μπορέσει η Κομισιόν να λάβει το Νοέμβριο απόφαση σχετικά και το πρόγραμμα θα μπορέσει έτσι να ξεκινήσει στις αρχές του 2019. Στόχος μας είναι το Διεθνές Κέντρο Μεταναστευτικής Πολιτικής ICMPD να είναι αυτό το οποίο θα αναλάβει τη διαχείριση. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στους βουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις, να κάνετε παρατηρήσεις. Λοιπόν, τώρα το λόγο έχουν οι βουλευτές. Okay, euh, Λοιπόν, ξεκινάμε με τους βουλευτές. Η κυρία Βεκαπέρα πρώτη. Έχετε το λόγο. Στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στο παρευρισκόμενο κοινό μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και θα σας δώσουμε το λόγο. Ξεκινάμε τους βουλευτές όμως. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω φιλανδικά, επομένως φορέστε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις που κάνατε και γιατί μας διαφωτίσατε πολύ περισσότερο για το ζήτημα αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ, ο οποίος έστειλε ένα πολύ χειρό μήνυμα, αναφέρθηκε στην Αφρική, αναφέρθηκε στη μετανάστευση και εν γέννη συμφωνώ μαζί του όταν λέει ότι θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερες εταιρικές σχέσεις και ότι θα πρέπει να καινοτομήσουμε, να ακούσουμε πολλές νέες ιδέες όσον αφορά την νέα αυτή μορφή αναπτυξιακής συνεργασίας. Ακούσαμε σήμερα από εσά πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν σε τοπικό επίπεδο. Ακούσαμε επίσης και ποια είναι τα εμπόδια και τα προβλήματα στην αναπτυξιακή συνεργασία. Νομίζω ότι θα πρέπει, όπω είπατε και εσείς, να αναφερθούμε σε κάποιε βασικέ υποδομέ όπω η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη. Είναι τομεί επί των οποίων χρειάζονται σαφώ περισσότερε επενδύσει, Και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν βέβαια και τα πιο παραδοσιακά μέσα αναπτυξιακή συνεργασία. Αν δούμε τι έχει γίνει πρόσφατα στον τομέα τη εκπαίδευση στι αναπτυσσόμενε χώρε. δεν είναι μόνο η πρόσβαση στην εκπαίδευση που αποτελεί πρόβλημα, αλλά και το παρεχόμενο επίπεδο εκπαίδευσης στις χώρες αυτές. Αν το συγκρίνουμε δηλαδή αυτό με το παρεχόμενο επίπεδο παιδείας σε ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει λοιπόν να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να συνεχίσουμε την παραδοσιακή αυτή αναπτυξιακή συνεργασία που, που είχαμε μέχρι τώρα ή αν θα πρέπει, όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ, να κινηθούμε προς ε, νέες μορφές συνεργασίας που θα περνάνε από τις επενδύσεις και κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης και σε πολλές άλλες περιοχές της Αφρικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος βουλευτής που θα θέλει να πάρει το λόγο. Νόρμπερτ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο γι' αυτό που είπε ο κύριος Στάουσμπολ πριν από λίγο, όταν μας είπε ότι αύριο θα ληφθεί μια απόφαση, ενδεχομένως από κοινού με τα κράτη-μέλη, προκειμένου να συσταθεί μια πλατφόρμα έτσι ώστε να δίδονται περισσότερες ευκαιρίες στους εκπροσώπους της Αφρικανικής Διασποράς, να μπορούν δηλαδή να επενδύουν μέσω της πλατφόρμας αυτής στις χώρες καταγωγής τους. Πώς θα γίνει αυτό στην πράξη. Είπατε κάτι για 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι δεν είναι. Αυτό είπατε στην αρχή της ε, παρέμβασής σας. Σας ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο μπορούν να πάρουν οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρίαση. Είχατε ζητήσει το λόγο. Κοίτα, ένα λεπτό, σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω για τα ζητήματα αυτά τα οποία αναπτύξατε. Είμαι ασκούμενη στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα απευθυνόμενη στον κύριο Ντόπ να το και μία ερώτηση. Από το Μαλή είμαι. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω όταν αναφέρεστε στον ρόλο της Αφρικανικής Διασποράς, είπατε ότι σαφώς μπορούμε να ενημερώσουμε περισσότερο τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές για την Αφρική. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι κατεστημένοι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κατάγονται από την Αφρική και θα μπορούσαν πραγματικά να καθοδηγήσουν τους υπεύθυνου για τη λήψη αποφάσεων. Νομίζω όμως ότι ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε και λίγο περισσότερο στους νέους που βρίσκονται εδώ πέρα στην Ευρώπη. Πώς μπορούμε δηλαδή να τους εμπλέξουμε και αυτούς περισσότερο, να φέρουμε στους νέους της Αφρικανικής Διασποράς. Πώς μπορούμε να τους κινητοποιήσουμε περισσότερο. Σας ευχαριστούμε. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση στην κυρία Μάνκε. και πείτε μας κι εσείς όμως ποιος είστε. από τη Διεθνή Ομάδα Περισυλλογής Προβληματισμού Αναφορά τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν στο Κονγκό. Θα ήθελα να γνωρίζω ποιους μηχανισμούς χρησιμοποιεί για να σε επαφή με μέλη της Αφρικανικής Διασποράς εδώ στην Ευρώπη και απευθυνόμενος επίσης και στον κύριο Στάσου Μπολ θα ήθελα να γνωρίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια μέσα διαθέτει στην Αφρικανική Διασπορά προκειμένου να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Σας ευχαριστούμε. Να υπενθυμίσω εδώ στο κοινό ότι ε, αν θέλετε να πάρετε το λόγο έχετε χρόνο αγόρευσης ε, ενό λεπτού. Τον έχετε τηρήσει περισσότερο μέχρι τώρα. Καλημέρα σα κυρία Κέγγε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Μαρή Πιέρνιε Τανί. Είμαι υπεύθυνη για την πολυμερή πλατφόρμα εκπροσώπησης των γυναικών τη Αφρικανικής Διασποράς. Μία παρατήρηση θα θέλω να κάνω. Θα ήθελα να μιλάμε για πολλές διαφορετικέ διασπορές και όχι για μία ενιαία διασπορά όπω την προσεγγίζουμε μέχρι τώρα. Η διασπορά έχει πολλές διαφορετικές πτυχές και το πρόβλημα είναι ότι ακριβώς επειδή είμαστε κατακαιρματισμένοι αυτή τη στιγμή, η δράση μας δεν είναι ιδιαίτερα ορατή. Απευθυνόμενοι στον κύριο Ντιόπ, θα έλεγα ότι υπάρχουν πρωτοβουλίε και στην Ευρώπη αλλά και στην Αφρική, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεταξύ μόνο κάποια επικοινωνία, κάποια διασύνδεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε τι κάνει κάθε πλευρά, ποιο κάνει τι και πώ μπορούμε τελικά να ομαδοποιήσουμε τι προσπάθειέ μα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, Μινώτα Κιντά από την Ρώμη. Ποιος είναι ο ρόλος της Αφρικανικής Διασποράς. Είπατε ότι η Αφρικανική Διασπορά μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε πάρα πολλές πτυχές. Έχουμε την Αφρικανική Διασπορά στην Ευρώπη, η οποία πολλές φορές βρίσκεται σε υποδέστερη θέση, όπως αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Λέμε από την άλλη ότι η Αφρικανική Διασπορά θα μπορούσε να εργαστεί και στην Αφρική και να συμβάλλει στην εκεί ανάπτυξη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έλλειψη ενημέρωση, ένα κενό ενημέρωση. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή από πού μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε, πώ μπορούμε να έχουμε μια υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναλάβουμε δράση στην Αφρικανική Ήπειρο. για όσους βρίσκονται στην Ευρώπη και ανήκουν στην Αφρικανική Διασπορά. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί που να, να μας επιτρέπουμε να γνωρίζουμε πόσοι είμαστε τελικά, πόσοι εργάζονται. Αυτή τη στιγμή η γενικότερη εντύπωση που υπάρχει στην Ιταλία είναι ότι περισσότεροι νέοι Αφρικανοί, μέλη της Αφρικανικής Διασποράς εκεί, δεν εργάζονται. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω αν έχουμε πιο αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά την κατάσταση της Αφρικανικής Διασποράς στην Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο διπλανός σας έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στα ισπανικά όμως θα τις κάνω. Επομένως φορέστε τα ακουστικά σας παρακαλώ πολύ, δεν καταλαβαίνετε ισπανικά. Λέγομαι Βένκα Κιέγκα. Είμαι πρόεδρος του Σάντρο Ευρωάφρικα, έτσι λέγεται η οργάνωση Μέτρα τη Βαρκελόνη. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την Σεσίλ Κιέγκε που μα απίφθινε πρόσκληση και βράτω με τι ευκαιρίε για να κάνω το εξή σχόλιο. Σε ό,τι αφορά τη διασπορά, το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό αλλά ταυτόχρονα με βάση την εμπειρία που έχω από την Ισπανία, πολλοί κόσμος ε, από τη Διασπορά δεν έχει πληροφορίες για το τι συμβαίνει, ας πούμε, εδώ στις Βρυξέλλες. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρχει μια ανταλλαγή και συνέργειες, γιατί το μεγάλο πρόβλημα, ιδίω στο Νότο ε, το εντοπίζουμε και είπε και η κυρία Κέγγε ότι τα προβλήματα ουσιαστικά είναι τα ίδια ε, που έχουν να κάνουν με τη μεταναστά. Τα τελευταία χρόνια όμως η Ισπανία ήταν μια χώρα διέλευσης, αλλά τώρα έχει γίνει μια χώρα υποδοχής. Ό,τι αφορά τους ανηλίκους, ε, είναι ένα πολύ ενσχετικό πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί ανήλικοι. Ε, ε, μιλώ κυρίως για την γαλλόφωνη Αφρική. Ε, πρέπει να το σκεφτούμε. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο μέρος που είναι αγγλόφωνο και πρέπει να δούμε εμείς τα μέλη της Διασποράς και εσείς που είστε εδώ, τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω να πω και κάτι ακόμη. Χαίρομαι που, πρέπει να, που αρχίζει να ασχολείται σοβαρά με το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει να ακούσει καλύτερα τη διασπορά. Είναι πολλοί αυτοί που ξέρουν πολύ καλά τα πράγματα. Μιλάω για την Ισπανία αλλά και για την Πορτογαλία και άλλες χώρες. Η διασπορά είχε μείνει εκτός της συζήτηση. Τώρα ε, αρχίζει να ακούγεται η φωνή της. Ε, πολλές φορές ξεκινάμε από το μηδέν. Πρέπει να πω όμω ότι, και το έλεγα για την Ισπανία που ξέρω, ο κόσμο που ξέρει και έχει πολλέ ε, γνώσει και μπορεί να προσφέρει πολλά είναι απογοητευμένοι γιατί έχουν μείνει στο περιθώριο. Είναι καλό λοιπόν η διασπορά να γίνει μέλο αυτή τη όλη προσπάθεια. Merci Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε τις ερωτήσεις στο σημείο αυτό για να δώσουμε τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Um, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κέντζε. Δεν έχουμε να κάνουμε εμείς παρατηρήσεις. Πολύ ωραία. Μόνο να προσθέσω κάτι όσον αφορά τα δίκτυα των νέων, όσον αφορά την Αφρικανική Διασπορά. Έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία με τρία τέτοια δίκτυα, Αντίνα, η ΦΥΣΕ και η FCPYN. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Στρέφουμε τώρα προς τους καλεσμένους μας. Θα θέλω να τους ξαναδώσω το λόγο για να απαντήσουν στις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις που ακούσαμε από τους βουλευτές και από τους συμμετέχοντες στη σημερινή συνεδρίαση. Η κυρία Μάγκη έχει πρώτη το λόγο. Σας δίνω μερικά λεπτά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις και σας υπενθυμίζω ότι έχουμε στη διάθεσή μας περίπου ένα τέταρτο, 15 λεπτά. Έχετε λοιπόν τρία λεπτά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, ερωτήσεις αλλά και ευχαριστώ τους ομιλητές που ήρθαν εδώ για να παρουσιάσουν τις εμπειρίες και τις πρωτοβουλίες τους. Ε, όλοι με το ίδιο θέμα ασχολούμαστε και θέλουμε να στείλουμε το ίδιο μήνυμα. Εταιρικές σχέσεις, συνεργασία, αποτελεσματικότητα, συμπληρωματικότητα και θεωρώ ότι ε, η ερώτηση της ε, Φιλανδίνας, ε, Φιλανδής Βουλευτίνας είναι πολύ σημαντική για τη χρηματοδότηση. Πώς βλέπουμε δηλαδή την επίπτωση επιτόπου στο πεδίο και πώς αντιμετωπίζουμε τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν πολύ τη χώρα προέλευσης. Οι επενδύσεις είναι σημαντικές. Χαίρομαι πολύ και ακούω με χαρά ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές επενδύσεις από τράπεζες και ιδιωτικό, από τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή για την, να διευκολυνθούν οι ροές των ε, χρημάτων. Όμως δεν είναι μόνο θέμα επενδύσεων, οικονομικών επενδύσεων. Υπάρχει και η επένδυση στην, ε, στους ανθρώπους, στην ε, ανάπτυξη τους. Εδώ μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο, γιατί μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο διαφορά. Αν χτιστεί ένα σχολείο, αλλά το ποιο θα πάει στο σχολείο είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε στο πόσο μπορεί η διασπορά να επιστρέψει ως μέντορες με συγκεκριμένους στόχους. Άρα, ναι, επενδύσεις σε δεξιότητες και στη δημιουργία δικτύων και δεξιοτήτων. Επίσης, ερώτηση πού υπάρχουν τα μέσα. Αυτή η ιδέα της πλατφόρμας της Διασπόρας όπου ανεβάζουμε όλες τις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, τα μενού που αναπτύξαμε, 150 χαρτογραφήσεις, όλα αυτά θα πάνε σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα γιατί θέλαμε και εμείς να ενημερωθούμε και φυσικά να ενημερώσουμε τους εταίρους. Ελπίζω λοιπόν ότι εκεί θα βρείτε πολλά. Φυσικά το πιο βασικό ε, είναι ένα εγχειρίδιο για την συμμετοχή, την εμπλοκή που συντάχθηκε σε ε, συνεργασία με τους εταίρους μας, το MPI και άλλους. Επίσης, η αφήγηση ήταν πολύ σημαντική και η γνώση για το τι ακριβώς κάνουν οι μετανάστες, γιατί συμφωνώ. Δεν υπάρχει μία διασπορά. Υπάρχουν άτομα ε, ε, από τη διασπορά και εγώ με διασπορά, ζω εκτός της χώρας μου επί χρόνια. Πολύ. Το θέμα είναι ποιος είναι σημαντικός όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα θεωρώ ότι έχετε δίκιο. Τα νούμερα, ναι, είναι 150, 280 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, είναι πολλά, αρκετά, λίγα, αλλά οι ιστορίες της διασποράς, τα χαρακτηριστικά τους είναι σημαντικά και γι' αυτό με την παρουσίασή μου έλπιζα να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα για τις επισκέψεις συγκεκριμένων, σε συγκεκριμένα χωριά που γίνονται συγκεκριμένα πράγματα, ας πούμε μια ε, μονάδα αλληλείας ή μια, ένα ε, εργοστάσιο θα σταματήσω εδώ γιατί από αυτόν ήθελα κυρίως να μιλήσω. Θα συνεχίσουμε να, τις συνομιλίες με τους ε, ομολόγους μας από την Κομισιόν και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ε, αλληλοσυμπληρωθούμε. Ευχαριστώ. Merci. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Λιόπ. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ε, σας ευχαριστώ. Θα συμπληρώσω αυτά που ακούστηκαν για το ρόλο των επενδύσεων και ποιο είναι το, η, ισορροπία μεταξύ επενδύσεων και κοινωνικής επένδυσης. Μιλάμε πολλές για επενδύσεις, αλλά ε, θέλουμε επενδύσεις με κοινωνικό αποτέλεσμα. Και ήθελα με αυτά τα παραδείγματα να φέρω αυτά με το ΡΑΣ, τα θέματα υγείας, παιδείας και πώς θα βοηθήσουμε τους νέους να αλλάξουν συμπεριφορά. Αυτή εδώ η συνεργασία η εταιρική σχέση είναι πολύ σημαντική γιατί συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως επίσης και με τα Ηνωμένα Έθνη και με το δημοσιοτικό τομέα. Εμείς είμαστε... Ε, δεν έχουμε μέσα που μπορούμε να μας επιτρέπουν να κάνουμε ταινίε, αλλά έχουμε εταίρους ε, και τηλεοπτικά κανάλια και λοιπά στη Γαλλία και στην αλλαγή αυτή της προσέγγισης όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον για το πώς μπορούν να ενισχυθεί η επίπτωση των επενδύσεων στην Αφρική. Ο καλύτερος τρόπος μείωσης της φτώχειας είναι η δημιουργία θέσεων εργασία, γι' αυτό χρειάζονται επενδύσεις και δημιουργία ε, προστιθέμενης αξίας. Επίσης, θέλω να απαντήσω στο, στην ερώτηση της κυρίας από το Μαλή αν κατάλαβα καλά, ότι πρέπει κανείς να πάει επιτόπου Δεν μπορεί να εκτιμήσει τις επιπτώσεις. Εγώ ήμουν στην Αφρική μέχρι το 2008. Επέστρεψα στη Σενεγάλη, όπου δημιούργησα μια εταιρεία μικροχρηματοδότησης με σκοπό την, ε, την δουλειά επιτόπου επέστρεψα στην Ευρώπη και φυσικά η ιδέα είναι η προσέγγιση να είναι κυκλική. Να μπορεί κανείς να πηγαίνει και στις δύο υπήρους. Να έχει από ένα πόδι σε κάθε μια για να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την εμπειρία και για την Ευρώπη και για την Αφρική. Και να συνεχίσει να εργάζεται με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα υπάρχουν μέσα επικοινωνίας φυσικά που μας επιτρέπουν να να δουλέψουμε σαν να ήμασταν εκεί. Μεσοπρόθεσμα η ιδέα είναι να ε, έχει κανείς παρουσία στην Αφρική. Αλλά δεν είναι ανταγωνισμό, ανταγωνιστικό το ένα με το άλλο. Αυτό που είπατε εσείς κύριε δεν ε, ε, έχω αντίρρηση αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε εκ των υστέρων το θέμα όσον αφορά τον συντονισμό και τον πολλαπλασιασμό των διαφορετικών πρωτοβουλίων, έχετε δίκιο. Εγώ θεωρώ σήμερα ότι πρέπει να σας παρουσιάσω με συγκεκριμένο παράδειγμα τι μπορεί να κάνει η διασπορά συγκεκριμένα και με βάση την εμπειρία μας πώς μπορούμε να προσφέρουμε για να αλλάξει η εικόνα της Υπήρου αλλά και να, εμπλακού, να εμπλακεί περισσότερο η διασπορά. Είμαι σίγουρος ότι η κυρία Μαρισοντάλ θα δώσει ε, πληροφορίες για τον τρόπο πώς μπορούν τα μέλη της Διασποράς να συντονιστούν για να δράσουν καλύτερα. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, euh, Monsieur Diop. Je... Σας ευχαριστώ κύριε Διόπ. Η Μαρία Σαντάλ, έχει τώρα το Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω στο ερώτημα για την κακή κατανόηση και το στιγματισμό ε, των ε, ανθρώπων. Πολύ σωστά το είπατε και ακριβώς γι' αυτό το λόγο η Παγκόσμια ημέρα διασποράς που οργανώνεται έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης για να καταλάβουν τι θα πει η διασπορά και τι προσφέρει η διασπορά. Εγώ είμαι στην Ιταλία και θέλω να σας πω ότι στο πλαίσιο της εβδομάδας ε, της Διασποράς ε, οργανώνονται στη Ρώμη εκδηλώσεις. 10 Οκτωβρίου συγκεκριμένα. Για να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία πληροφορικής, τεχνολογιών, ε, επικοινωνιών πληροφοριών, για να καταπολεμήσουμε ακριβώς τη στιγματοποίηση. Και κάτι άλλο που θέλω να πω είναι να στηρίξω το μήνυμα της βουλευτού για την ανάγκη να ξαναδούμε την εταιρική σχέση μεταξύ Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι, μπορεί να μην ακολουθήσει η Αφρική το ίδιο ε, μονοπάτι με την Ευρώπη, την ίδια διαδρομή. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο, ποιε είναι οι τοπικέ ανάγκες. Σήμερα στην Αφρική υπάρχουν πραγματικές ανάγκε σε θέσει εργασία. Χρειάζεται εκβιομηχάνηση, αξιοποίηση των φυσικών πόρων για την ανάπτυξη της αφρικανικής οικονομίας. Και νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες, γιατί αυτό σημαίνει θα πρέπει να υιοθετήσουμε αποτελεσματικέ πολιτικές. Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση άκουσα και εγώ την ομιλία του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ που είπε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να προσαρμοστεί στην εξέλιξη της Αφρικής και να συνοδεύσει την Αφρική σε αυτή την προσπάθεια και όχι να επιβάλλει στην Αφρική αυτό που θέλει έχουμε στις εταιρικέ σχέσεις και στην αποφυγή αλληλεπικαλύψεων. Πράγματι, είμαστε πολύ άριθμοι. Και όταν είμαστε πολύ άριθμοι, έχουμε την τάση ο καθένας να κοιτάει τα πράγματα από τη δική του οπτική και καλό θα ήταν να δείξουμε μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Και αν πηγαίνουμε στην ίδια κατεύθυνση, καλό είναι αντί να είμαστε διασπαρμένοι να ενώνουμε τι προσπάθειε και να μην υπάρχει αλληλεπικάλυψη. Αυτό είναι καλό και για το λέμε και στο διάλογο που κάνουν τις δημόσιε αρχέ. Γιατί πολλές φορές επειδή είμαστε πολλοί δεν ξέρουμε πού να απευθυνθούμε. Όσο πιο καλά οργανωθούμε, τόσο πιο καλά δομημένο θα είναι ο διάλογο και, και τόσο πιο αποτελεσματικό. πρόσωπος Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπα κάποια πράγματα. Εμεί είχαμε αναλάβει την πρωτοβουλία μαζί με την Κομισιόν να διοργανώσουμε μία ημερίδα μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διασποράς. Είμαστε ένας φορέας ανάπτυξης με μεγάλες ιδιαιτερότητες ως κοινό των πολιτών ε, δεν μπορούμε να μπούμε στο ίδιο τσουβάλι με όλους. Πρέπει να υπάρχει διάλογους. Τέτοιου είδους ε, εκδηλώσεις πρέπει να είναι κάτι που θα γίνεται συχνά και στο Κοινοβούλιο αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξού και η σημασία νομίζω να δημιουργηθεί μια συνεργατική πλατφόρμα διαβούλευσης όπου τα μέλη, οργανώσεις, ε, αντιπροσωπευτικές της διασπάρας θα μπορούν να ε, συναντώνται και να εξηγούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Και για να ολοκληρώσω, Θέλω να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση του μέσου για τη διασπορά, Facility for Diaspora. Και ελπίζω και οι αρχηγοί, μάλλον οι εκπρόσωποι των ε, κρατών, να ψηφίσουν, να ε, εγκρίνουν αυτό το σχέδιο για τις πρωτοβουλίες αυτές που θα ενισχύσουν ε, τη χρηματοδότηση Τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και ελπίζω επίσης να υποστηριχθούν πρωτοβουλίε που στόχο κυρίως θα έχουν την ένταξη των ε, ανθρώπων τη διασπορά, στις χώρε υποδοχή. Γιατί αν η διασπορά δεν έχει αγοραστική δύναμη, δεν μπορεί να στηρίξει και τις χώρε καταγωγή. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Στάουσμπολ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα θετικά σχόλια τα οποία κάνατε. Δεν το συνηθίζουμε πάρα πολύ εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούμε τόσο θετικά λόγια. Και ξέρετε ότι εδώ πέρα βασιστήκαμε πάρα πολύ στις βασικές αρχές της διαφάνειας, προσπαθώντας να σας ενημερώσουμε πλήρως για τα συστήματα υποστήριξης που υπάρχουν, ιδίως όσον αφορά την χρηματοδότηση. Πολύ σύντομα όσον αφορά τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, από την ε, κυρία Δεκαπέρα. Αυτό το οποίο ανακοινώσαμε τελικά πριν από δύο εβδομάδες, ε, τις δύο αυτές ανακοινώσεις όσον αφορά την Συμμαχία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Μέρος της απάντησης μόνο θα είναι αυτό. Κανεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση δεν έχει την ψευδέστηση ότι θα μπορούσαμε να καλύψουμε όλα τα αναπτυξιακά προβλήματα που υπάρχουν στην Αφρική μέσω των δύο αυτών ανακοινώσεων. Θέλουμε εμεί να ενισχύσουμε περισσότερο τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και θα πρέπει να δούμε εδώ πέρα πώς θα καταφέρουμε να σταθμίσουμε τη συμμετοχή των διαφορετικών φορέων για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το νέο ενιαίο μηχανισμό χρηματοδότησης, ο οποίος εφόσον εγκριθεί θα μπορέσει να συμβάλλει στην ε, ε, γενικότερη χρηματοδότηση. Ο κύριος Νόιζερ, εν συνεχεία, να διευκρινίσω δύο πράγματα είπα. Πρώτον, ότι ε, στα πλαίσια του του μηχανισμού εγγύησης 1,5 ε, εκατομμυρίου. Έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν ε, επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου της Αφρικανικής Διασποράς στην Αφρική και αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου αλλά είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αυτοί που θα διαχειριστούν τα ποσά αυτά και αν δείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήδη εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για το ποιοι είναι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που θα διαχειριστούν την, το μηχανισμό αυτοδιευκόλυνσης της χρηματοδότησης. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αναφέρθηκα σε ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο, το οποίο ελπίζω ότι θα εγκρίνουν αύριο στην Επιτροπή DCI τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι το ετήσιο πρόγραμμα 2018 για την ε, μετανάστευση στα πλαίσια του ε, πολιετούς προγράμματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα που θα έχει να κάνει με την ε, μετανάστευση από την Αφρική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σας είπα, δίνονται νέες δυνατότητες, υπάρχει ένα υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας. Ο αγαπητός συνάδελφος ε, που ασχολείται με την Αφρικανική Διασπορά και πήρε το λόγο πριν από λίγο, αναφέρθηκε και αυτός στα σημεία αυτά. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί καλεσμένοι, σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας, για τη συμμετοχή σας, για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Προετοιμάζοντας την ακρόαση αυτή, και στην εισαγωγική μου παρέμβαση είπα ότι θα πρέπει να εμπλέξουμε περισσότερο την αφρικανική διασπορά που βρίσκεται στην Ευρώπη, να την εμπλέξουμε περισσότερο στην αναπτυξιακή μας συνεργασία με την Αφρική. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, απευθυνόμενοι και στους βουλευτές αλλά και στο παρευρισκόμενο κοινό. Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε σε, στην καλύτερη δυνατή θέση για να ενισχύσουμε περισσότερο τη συμμετοχή της Αφρικανικής Διασποράς στην Ευρώπη για την πρόθεση αποτελεσματικών πολιτικών αναπτυξιακής συνεργασίας. Θα προσπαθήσω εντάχει να συνοψίσω την ακρόασή μας αυτή να αναφερθώ σε κάποια σημαντικά σημεία, σημαντικά συμπεράσματα. Ξέρουμε ότι η Αφρικανική Διασπορά απαριθμεί, πολύ, απαριθμεί περίπου 30 χρόνια και έχουμε πάρα πολλούς άνδρες και γυναίκες που συμμετέχουν σε αυτή την Αφρικανική Διασπορά και αυτή τη στιγμή δεν έχει να κάνει μόνο με μετανάστες οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα για οικογενειακού λόγους, αλλά και μετανάστες που έρχονται για οικονομικούς λόγους. Έχουμε πλέον και φοιτητέ και ειδικευμένου εργάτες Νέου επίση που έρχονται να σπουδάσουν, γυναίκε επίση ε, που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω τη εργασία θέλουν να υποστηρίξουν τι οικογένειε του. Ξέρουμε ότι διπλασιάστηκε τα 20 τελευταία χρόνια ο αριθμό των ε, Αφρικανικών μεταναστών με 9 εκατομμύρια που φτάσανε μεταξύ του 2000 και του 2017. Και 19 εκατομμύρια είναι συνολικά οι μετανάστες οι οποίοι φύγαν από τη χώρα καταγωγής τους στην Αφρική για να πάνε σε άλλες αφρικανικές χώρες. Η κυρία Μάνκε το ανέφερε και αυτό πριν από λίγο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Αφρικανοί οι οποίοι εγκαταλείπουν τις χώρες του Μαγκρέπ και την υποσαχάρη Αφρική για να έρθουν στην Ευρώπη. Όσοι έρχονται από την υποσαχάρη Αφρική και πηγαίνουν προς τη Γαλλία, την Ιταλία, τον Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτογαλία, προέρχονται κυρίως από την Ιγυρία, την Νότια Αφρική, τη Σομαλία, τη Σενεγάλη, την Γκάνα, την Αγγόλα, την Κένια, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, από το Καμερούν και προέρχονται επίσης και από την ακτή του Ελεφαντοστού. Συνοψίζοντα λοιπόν αυτά που μα είπε και η, Μαρία, κυρία Μαρίνα Μάνκε, έχουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα τα θα σα δώσουμε μέσα στι επόμενε μέρε. Αναφερθήκαμε επίση στο ζήτημα των εμβασμάτων. Τα εμβάσματα αυτά τα οποία φτάνουν σε ένα πολύ υψηλό ποσό, το οποίο υπερβαίνει την ε, επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Ο κύριο Τζόμπα αναφέρθηκε σε 65 εκατομμύρια ε, δολάρια το 2015, ενώ 50 εκατομμύρια δολάρια είναι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ποσού αυτού πηγαίνει στην υποσαχάρια Αφρική και τα εμβάσματα αυτά φτάνουν τα 9,3% του συνολικού ποσού όσον αφορά την υποσαχάρη Αφρική. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι τα δεδομένα αυτά ότι πρέπει να μιλάω πιο αργά για να με παρακολουθούν οι Είμαι πεπισμένη πάντως ότι παρακολουθήσατε ήδη πολύ καλά όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία μα παρουσίασαν οι παρεμβαίνοντε. Έλεγα λοιπόν ότι οι μετανάστες θα μπορούσαν να βοηθήσουν του επιχειρηματίε και του παραγωγού τη χώρα καταγωγή του να βρουν αγοραστέ στην Ευρώπη και θα πρέπει βέβαια να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν πλατφόρμες και φόρουμ. Αναφερθήκαμε και στις δυνατότητες αυτές και όλοι οι παρεμβαίνοντε άγγιξαν και το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά τώρα το ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και το παγκόσμιο επίπεδο, βλέπουμε ότι είδαμε μάλλον μέσω των παρουσιάσεων αυτών ότι δίνεται πάρα πολύ μεγάλη σημασία στον ρόλο που θα μπορούσε να έχει η Αφρικανική Διασπορά όσον αφορά μια τακτική μετανάστευση που θα γίνεται βάση των κανόνων. Ξέρετε ότι ήδη ε, τον Δεκέμβριο προβλέπεται μια συνεδρίαση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρικανική Ένωση για το Παγκόσμιο Σύμφωνο όσον αφορά τη μετανάστευση. Η διεθνή λοιπόν αυτή μετανάστευση είναι ένα σημαντικό ζήτημα και συνάδει επίσης και με τον στόχο 19 να δημιουργηθούν δηλαδή κατάλληλες συνθήκες προκειμένου οι διασπορά και μετανάστες να μπορούν να συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη παγκοσμίω. Ακούσαμε την κυρία Μαρή Σοντάλ Ουβιτονζέ, καθώ επίση και την παρουσίαση του κυρίου Ντιόπα και μέσω των παρουσιάσεών του βλέπουμε ότι οι στόχοι αυτοί ήδη έχουν αρχίσει να υλοποιούνται. Πρέπει παρόλα αυτά να τονίσουμε ότι η δράση της διασποράς έχει ένα πολυτομεακό χαρακτήρα όσον αφορά τα μέσα, τις στρατηγικές και τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν να κάνουν με την Αφρικανική διασπορά είδαμε μέσω των παρουσιάσεων κυρίως του κυρίου Σταουσμπολ ότι διαθέτουμε ήδη μια πολύ μεγάλη γκάμα μέσων που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Πολλές φορές όμως δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιο μέσο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει κοινή στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης, υπάρχει το Παναφρικανικό Πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το αναπτυξιακό μέσο του DSE, που έχει ως στόχο να δυναμώσει περισσότερο τη συμβολή της διασποράς για την ανάπτυξη της Αφρικής. Προβλέπεται επίσης η πρόθεση του διαλόγου για τη μετανάστευση και την κινητικότητα. Η συμβολή λοιπόν της διασποράς όσον αφορά την ανάπτυξη των χωρών καταγωγής καλύπτεται όπως βλέπετε και από άλλα μέσα. Ακούσαμε επίσης να γίνεται αναφορά σε ένα πρόγραμμα του DCI το οποίο θα παρουσιαστεί πολύ σύντομα και το οποίο ουσιαστικά έχει ως στόχο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ε, παγκόσμιες προκλήσεις ε, που ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσει παγκοσμίως η αφρικανική διασπορά. Μέσω του προγράμματος αυτού θα δοθούν 5 εκατομμύρια, 5 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποσαχάρη Αφρική συγκεκριμένα. Είναι πολύ σημαντικό επίση να ασχοληθούμε με το ζήτημα των εμβασμάτων, ζήτημα με το οποίο ήδη καταπιάνεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Τα εμβάσματα αυτά θα πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικά, να έχουν ε, θετικέ, γρήγορε επιπτώσει για την αγορά τη Αφρική. Θα πρέπει λοιπόν να χαιρετήσουμε τι νέε αυτέ πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση όσον αφορά τα εμβάσματα. Θα ήθελα πολύ γρήγορα να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα, γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε και με τι ψηφοφορίε μα. Εν κατακλείδη λοιπόν θα έλεγα ότι α, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων απέναντι σε όλους τους καλεσμένους μας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους. Η Επιτροπή μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς ε, το ζήτημα αυτό και να υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που θα έχει ως στόχο να προωθήσει περισσότερο τη συμμετοχή της Αφρικανικής Διασποράς στην Ευρώπη για την προώθηση αποτελεσματικών πολιτικών αναπτυξιακής συνεργασίας στην Αφρικανική Ήπειρο. Σα ευχαριστώ. Je rappelle... Σας υπενθυμίζω, υπενθυμίζω στα μέλη ότι η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 5 παρατέταρτο, ακριβώς 9 λεπτά δηλαδή. Okay, ladies Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ καθίστε για να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία που προβλέπει η συνεδρίασή μας. Καθίστε. We will start θα ξεκινήσουμε από τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές στη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Έχουμε τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Θα αρχίσει τώρα η ψηφοφορία, αν είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι όλοι. Πρώτο, συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος, έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν. Μετά, η 26, τροπολογία 26, περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται θα πω, <laughs> ναι. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32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 αποχές, κατά, αποχές, Ας ελέγξουμε. 38, έλεγχος για τη 38. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 46 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 50. Υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατόπιν η συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατόπιν συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 ε, λέει η πρόεδρος, όχι, 56 λοιπόν, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατόπιν θα ψηφίσουμε για την 57, αλλά θα γίνει χωριστή ψηφοφορία σε τρία μέρη, ενώ το τέταρτο μέρος αφαιρείται. Θα ψηφίσουμε επί των τριών μερών. Πρώτο, ξεκινώντας από το no later than μέχρι το ε, outside the union, και μετά and every two years thereafter. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Ψηφίζουμε για το πρώτο μέρος λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος ε, αφορά τον όρο those words. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το τρίτο μέρος αφορά το σημείο It shall also evaluate the contribution και the Commission may present appropriate legislative proposals. Αυτό Ψηφίζουμε υπέρ του τρίτου. Κατά αποχές εγκρίνεται. We move to aim 9. Περνάμε κατόπιν στην τροπολογία παριθμών 9. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. η 10. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η δεκατέσσερα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική δύο Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ή 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κατόπιν έχουμε τη συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας κάνουμε έλεγχο. Για την 19. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Έχουμε τώρα μια τελική ψηφοφορία επί του συνόλου της, του σχεδίου γνωμοδότησης και θα χρησιμοποιήσουμε το μηχάνημα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 11 υπέρ και μία κατά. 5 αποχές. Αυτά. Σχετικά με το μέρος αυτό, κατόπιν προχωράμε στο δεύτερο κατάλογο ψηφοφοριών 24η διάσκεψη των μερών της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Θα δώσουμε καταρχήν το λόγο Μαρσέλες, το Μαρσέλες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να επισύρω την προσοχή των συναδέλφων στην παράγραφο 8 διότι εντυπωσιαστήκαμε ε, ξεπλάγημεν για το συμβιβαστική επί της ε, παραγράφου 6, ενώ πριν από δύο εβδομάδες ψηφίστηκε μια θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην παράγραφο αυτή δεν αναφέρεται η θέση αυτή που ψηφίστηκε στο Στρασβούργο. Άρα η τροπολογία των πρασίνων είναι, έχει σκοπό απλώς να αποκαταστήσει αυτό που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία προ δύο εβδομάδων. Απλώς αυτό. Okay, then we vote number. Λοιπόν, η τροπολογία παριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κατόπιν, τροπολογία υπαριθμών 2, λέει η ε, πρόεδρος, που χωριστεί ψηφοφορία σε τρία μέρη. Συγγνώμη. Αν είπα κάτι άλλο, εννοούσα τρία. Τροπολογία υπαριθμών 3, λέει η πρόεδρος. Λοιπόν, τροπολογία υπαριθμών 3. Ψηφίζουμε ε, σε δύο μέρη. Πρώτον, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, ε, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας, απορρίπτεται. Το δεύτερο μέρος, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα, υπαριθμόν τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και κατόπιν η έξι υπέρ κατά αποχές ας κάνουμε έναν έλεγχο της έξι έναρξη ψηφοφορίας πέρας εγκρίνεται τελική ψηφοφορία επί του συνόλου ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 12 ψήφους υπέρ, 5 κατά και μία αποχή. τα πήγαμε αρκετά καλά νομίζω στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ πολύ όλους. Okay.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 συνεχίσουμε. Καθίστε παρακαλώ. Έχουμε τώρα την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σε σχέση με την απόφαση σύνδεσης υπερπόντιων χωρών εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ρυθμίζει τις μελλοντικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ε, υπερπότιες χώρες και δάφη και την Γρυλανδία. Όπως προβλέπεται στη διαδικασία διαβούλευσης, θα πρέπει το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν λάβει απόφαση. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο μόλις ξεκίνησαν, επομένως είναι επίκαιρη αυτή η πρώτη γενική ανταλλαγή απόψεων που οργανώνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου θα υποβληθεί από την ε, Κομισιόν. Επίσης έχουμε καλέσει τον Κάρολ Βόγκες, πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής ε, της ε, Ένωσης των Περπόντων Χωρών και Εδαφών, ΟΚΤΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος αυτής της Ένωσης είναι συλλογική εργασία με την πρόθεση κοινών θέσεων και εταιρικών σχέσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη των ΙΧΕ. Δεύτερη θητεία. ενός έτους διάρκειας το Φεβρουάριο 18 για τον Κάρολ Βόγκης. Δυστυχώς δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ η συγγητής μας, ο Μωρής Πονγκά. Θα αντικατασταθεί από την κυρία Ζηλιάνα Ζόφκο. Καταρχάς η Σιλβή Μιλό θα πάρει το λόγο, που είναι η τμήματάρχης από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ για θέματα που άπτονται τον ε, ΙΧΕ. Περπόντων χώρων και να Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ που μπορώ να σας παρουσιάσω την πρόταση της Κομισιόν για τη νέα απόφαση περί σύνδεσης Ευρωπαϊκή Ένωση. και μια ευκαιρία για να σας συστηθώ Λέγομαι Σιλβί Μιγιό, είμαι νέα τμήματάρχης, αρμόδια για τι σχέσει με τι ε, ΙΧΕ, στη γάμα δέλτα ντεύκο τη Κομισιόν. Τρεις εβδομάδες πάει που ανέλαβα τα νέα μου καθήκοντα και ελπίζω να έχουμε επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και σήμερα και στο μέλλον. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες γενικές πληροφορίες για να σας παρουσιάσω τα ΙΧΕ που είναι 25 σε σχέση με 4 κρατη κράτη-μέλη, Γαλλία, Ολλανδία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο. Με μεγάλη πολιτική σημασία για τα κράτη-μέλη αυτά βέβαια, αλλά και για την Ένωση συνολικά. Όλα τα ηχεία είναι νησιά, από το τροπικό μέχρι ε, τους πόλους, μικρά σε μέγεθος ε, και με αραιό πληθυσμό. Και όλα έχουν πολύ μεγάλο ρόλο να δραματίσουν σε διάφορες περιοχές ε, της Ένωσης αλλά και άλλων περιοχών Καραϊβική, Ειρηνικός ε, μέχρι την Αρκτική, Ανταρκτική με μεγάλη αυτονομία σε τομείς όπως οικονομικές υποθέσεις, απασχόληση, δημόσια υγεία, εσωτερικά ζητήματα, τελωνιακά ζητήματα και όπως και οι άκρως απόκεντρες περιφέρειες δεν εντάσσονται στη, μάλλον αντίθετα από τις απόκεντρες δεν εντάσσονται στην αγορά, ούτε στην ενή αγορά, ούτε δεσμεύονται από το κοινοτικό κεκτημένο. Όμως από την αρχή ήταν μέλος της οικογένειας της Ένωσης, γιατί υπήρχε συμφωνία σύνδεσης από τότε που τέθηκε σε ισχύ συνθήκη της Ρώμης. Okay. So why a new decision Γιατί μια νέα πρόταση απόφασης. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο αποφάσεις σε σχέση με τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ΙΧΕ. Πρώτον, την απόφαση περί σύνδεσης, η οποία εγκρίθηκε το 2013 και δεν έχει καταληκτική ημερομηνία. Και δεύτερον, η απόφαση για τη Γρυλανδία που εγκρίθηκε το 2014 και θα λήξει το 2020. Πρέπει να πούμε ότι η Γρυλανδία καλύπτεται από την απόφαση περί σύνδεσης. βασικός λόγος για να έχουμε μια επιπλέον απόφαση είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι η μόνη χεία που χρηματοδοτείται από τον Ενωσιακό Προεπολισμό. Οι άλλε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη χρηματοδοτούνται. Γιατί θέλουμε να συγχωνεύσουμε αυτέ τώρα τι δύο αποφάσει. Πρόταση είναι αυτό να γίνει, να συγχωνευτούν αυτές οι δύο αποφάσεις και αυτό ε, για διάφορους λόγους. Θέλουμε καταρχάς να απλουστεύσουμε και να ενοποιήσουμε τα εξωτερικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με μία ενιαία απόφαση για όλα τα είχε. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τους, με τους στόχους μας. Δεύτερον, το Brexit. Τέλη Μαρτίου του 2019 υπολογίζουμε το Brexit. Δεν θα καλύπτεται λοιπόν το Brexit με αυτή την απόφαση. Για Γαλλία, Δανία και Ολλανδία πλέον θα ισχύουν μόνο. Και επίσης ε, η εγγραφή του ΕΤΑ στον προπολογισμό και οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχει νέα γραμμή στο 6, στην κατηγορία 6 για τη γειτονία και τον κόσμο. Νέος λοιπόν προϋπολογισμός, νέα γραμμή προϋπολογισμού. Ήταν κάτι που το είχε ζητήσει στο Κοινοβούλιο. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης. Γενική αρχή. Ποια είναι η προσέγγιση πρότασης. Να διατηρηθεί αυτό που λειτουργεί καλά. Ο στόχος και τα βασικά χαρακτηριστικά της ε, ένωσης παραμένουν. Τη σύνδεση, συγγνώμη. Η δομή παραμένει ίδια. Επικαιροποιείται το περιεχόμενο για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις από το 2013 ορισμένους και καταργούνται τα απαρχαιωμένα στοιχεία. Καλύπτονται τα θέματα που έχουν να κάνουν με εμπορικές πολιτικές ε, σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ ΙΧΕ και Ένωσης, ορίζονται οι κατευθυντήριε γραμμές και οι φορεί πολιτικού διαλόγου. Μεταξύ κρατών μελών, ΙΧΕ και Ένωσης τομείς δράσης, ε, τα οικονομικά ζητήματα και οι εμπορικέ διευθετήσεις. Περιλαμβάνονται επίσης ειδικέ διατάξεις ε, όταν αυτό είναι απαραίτητο, οι οποίες συγκεκριμένα θα διέπουν την εταιρική σχέση με τη Γρυλανδία. Οι ΧΕ παραμένουν επιλέξιμα για τα προγράμματα της Ένωσης, αυτό παραμένει αρχή, εκτός αν δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Για να μην υπάρχουν παρανοήσεις στο μέλλον, τα προγράμματα της Ένωσης θα αναφέρω συγκεκριμένα το αν είναι δυνατόν υπάρχει επιλεξιμότητα για τις ε, περπόντε χώρε και ταυτή. Αλλάζει λοιπόν εν σύντομη. Τώρα προτείνουμε μια νέα απόφαση που καλύπτει 13 είχε χωρί ε, τα 12 που έχουν να κάνουν με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα έχουμε έναν προπολογισμό. 500 εκατομμύρια ευρώ είναι το προτινόμενο ποσό για τα ΙΧΕ στο πλαίσιο του νέου πολιτισμού συνομικού πλαισίου. Ένα ποσό το οποίο ε, το έχουμε αφαιρώντας ε, τις, ε, τα κεφάλαια που πήγαιναν ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουμε αύξηση 3,3% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Για να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για το ποσό αυτό, 225 εκατομμύρια πάνε στην Γρυλανδία και 225 στα άλλα 12 είχε. Από το τελευταίο αυτό ποσό, 159 εκατομμύρια θα δοθούν σε εδαφικά προγράμματα, δηλαδή διμερή συνεργασία και 81 εκατομμύρια για περιφερειακά προγράμματα. Και εδώ κάτι καινούργιο έχουμε ειδικό κονδύλι για την διαπεριφερειακή συνεργασία. Επίσης, 22 εκατομμύρια προβλέπονται για μελέτες. Στήριξη στην Ένωση ε, της, ε, τη συμφωνία μάλλον σύνδεσης και άλλοι. Και 13 εκατομμύρια για πρόβλεπτα, για στάθμη τους, ε, για καταστάσεις, από θεματικό. Επίσης, ενισχύεται με την πρόταση η διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των ΙΧΕ, με τους γείτονέ τους. Υπάρχει το συγκεκριμένο κονδύλο που προανέφερα. Προβλέπεται η περιφερειακή συνεργασία με άλλες ΙΧΕ, με τις χώρες ΑΚΕ και τρίτες χώρες. Προστίθεται και η έννοια εδάφη, territories, για να υπάρχει δυνατότητα περιφερειακής συνεργασίας με τα εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου, που ήταν μια επίσης ανησυχία που είχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, κατάλογος των μεών συνεργασίας έχει προσαρμοστεί ελαφρώς για να λάβει υπόψη να τομείς που προηγουμένως ήταν μόνο στην απόφαση για τη Γρυλανδία, όπως ε, τα θέματα που έχουν την αρκτική, τις πρώτες ασφάλεια και φοδιασμό τροφίμων. Αυτές οι διατάξεις βέβαια θα εφαρμόζονται πλέον σε όλα τα ΙΧΕ, εφόσον η απόφαση συνολικά εφαρμόζεται σε όλα αυτά τα εδάφη. Ποιος είναι ο σύνδεσμος ε, λοιπόν με τις διαπραγματεύσεις ε, για το NDCI και το νέο πρόγραμμα. Υπάρχει σχέση. Το τελικό ποσό θα εξαρτάται από το τι θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές. Επίσης, στα θεματικά και τις διάφορες ενέργειες του NDICI θα είναι επιλέξιμα τα ηχεία και θα παραμείνουν επιλέξιμα και για το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, αν δεν λέγεται κάτι διαφορετικά, στη νέα αυτή συμφωνία σύνδεσης ε, θα εφαρμόζονται και οι κανόνες εφαρμογής ε, του DICI. Αλλά αν είναι αναγκαίο θα, και το ενθαρρύνουμε αυτό, θα προβλέπονται απλουστευμένοι κανόνες για τον προγραμματισμό, για παράδειγμα, μεταξύ άλλων. Για να ολοκληρώσω, έχουμε δύο γενικούς στόχους στους οποίους θέλει να επιτύχει αυτό το νέο σχέδιο απόφαση. Πρώτον, θέλουμε να λάβουμε υπόψη τι ιδιαιτερότητες ε, των υπερπόντιων ε, χωρών και δαφών αλλά ταυτόχρονα να παγιώσουμε και να διατηρήσουμε αυτό που λειτουργεί καλά. Θέλουμε να διατηρήσουμε επίση τι συνέργειε με άλλα εξωτερικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Και ο δεύτερο στόχο είναι να δοθεί μεγαλύτερη διαφάνεια, μάλλον μεγαλύτερη ορατότητα στο ειδικό καθεστώ των ΙΧΕ, με υψηλότερη προβολή ω ομάδα και ω τμήμα τη Ευρωπαϊκή Οικονομία. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και παραμένω στη διάθεσή σα για οποιοδήποτε σχόλιο και για να έχουμε μια συζήτηση. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ, Σίλβια. Ας ακούσουμε τώρα τον Κάρολ Βόγγες, την Κάρολ Βόγγες, η οποία είναι πρόεδρος της ε, Ένωσης ε, Υπερπόντιων Χωρών και Δαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτής της Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Κάρολ Βόγκε και είμαι πρόεδρο Εκτελεστική Επιτροπή τη Ένωση Υπερπότων Χωρών και Δαφών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόσκληση αυτή και τη δυνατότητα που μα δίνει να παρουσιάσουμε τη δική μα τοποθέτηση όσον αφορά την απόφαση και τη σύνδεση των υπερπόντων χωρών και δαφών. να σας κάνω μια σύντομη ιστορική αναδρομή της Ένωσής μας η πρώτη διάσκεψη έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2000, όπου είχαμε τότε την πρώτη κοινή μας θέση στα πλαίσια της 7ης απόφασης για τη σύνδεση των ΙΧΕ. Στην υπουργική διάσκεψη που έλαβε χώρα το 2002, δημιουργήθηκε η ΟΚΤΑ ως μη κερδοσκοπική οργάνωση με βάση το βελγικό δίκαιο και όπως υπόθηκε από την κυρία Μιλό, έχουμε 25 OCTs και έχουμε ε, τις ε, υπερπόντια εδάφη, τις υπερπόντιες χώρες από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες ε, δεν εκπροσωπούνται. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι παγκόσμια η παρουσία μας. Βλέπετε εδώ πέρα την δομή, τη διάρθρωση της Ένωσης. Έχουμε την Υπουργική Διάσκεψη, που είναι η ανώτερη υψηλόβαθμη μορφή λήψη αποφάσεων. Έχουμε επίση και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Έχουμε εκπροσώπηση από τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη. Συνεδριάζει η διάσκεψη αυτή σε αιτήσια βάση, θέτει τις προτεραιότητες για το επερχόμενο έτος. Η Γαλλική Πολυνησία αυτή τη στιγμή έχει την Προεδρία μέχρι την επόμενη συνεδρίαση και υπάρχει και μια εκτελεστική επιτροπή, στόχος της οποίας είναι η χειριστή της καθημερινές δράσεις της Ένωσης. Έχουμε και μια γραμματεία που παρτίζεται από τρία μέλη και επικεφαλής είναι συντονιστής, ο οποίος ε, είναι επικεφαλής επίσης και της ε, όλης επικοινωνίας και ενημέρωσης. Αυτή τη στιγμή ε, συζητάμε την πρόταση της ένατης απόφασης για τη σύνδεση των ΙΧΕ τον ε, Φεβρουάριο. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη μελλοντική εταιρική σχέση μετά το 2020 Είχαμε πρώτα την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο και εμεί αμέσως δώσαμε την άποψή μας σε σχέση με την ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης. Βέβαια δεν εκφράζει τοποθέτησή μας αυτή τις απόψεις της Γρυλανδίας. Στόχος μας και επιθυμία μας ήταν να διατηρήσουμε το κεκτημένο της υφιστάμενης απόφασης για τη σύνδεση των ΙΧΕ, να κρατήσουμε όλα αυτά τα οποία λειτουργούν καλά, να βελτιώσουμε όσα δεν έχουν λειτουργήσει καλά, όσον αφορά τους στρατηγικούς προσανατολισμούς. Η τελευταία απόφαση την οποία αναλύσαμε ήταν αυτή του 2009 και έγινε μια επικαιροποίηση εν συνεχεία το 2012 και το 2017. Είχαμε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμβαθύνει περισσότερο το όραμά τη και το στρατηγικό τη προσανατολισμό όσον αφορά την εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και υπερπόντων χωρών και εδαφών. Είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερε δυνατότητε διαλόγου στα πλαίσια τη υφιστάμενη απόφαση για τη σύνδεση των ΙΧΕ. Υπάρχουν διάφορα μέσα διαλόγου, ε, διάφορα μέσα διαβούλευση, ε, σύμφωνα με το άρθρο 14 του OAD Επίσης ε, έχουμε τις, ε, τα συμπεράσματα της 14ης, 15ης και 16ης συνεδρίασης Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερπόντων χωρών και εδαφών, όπου ε, προβλέπονται συστάσεις για την απόφαση του 16, του 17 και 18. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβλέπονται άνω των τριών ετησίων δυνατοτήτων για περαιτέρω διάλογο και διαβούλευση και μεγαλύτερη συμμετοχή και πιο δραστήριο ρόλο για τις υπερπόδιες χώρες και υπερπόντια εδάφη. Όσον αφορά τώρα την χρηματοοικονομική υποστήριξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις με ανώτατο ποσοστό 26%, αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι ο τοπικός αντίκτυπος ήταν μόνο της τάξης του 3,2%. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε άμεση χρηματοδότηση οι, τα υπερπόντια, οι υπερπόντιες χώρες, τα υπερπόντια θα θέλανε να διατηρηθεί το εφιστάμενο επίπεδο χρηματοδότησης και να μην μειωθεί αυτό με την νέα απόφαση. Να σας εξηγήσω τώρα πολύ γρήγορα πώς άλλαξαν διάφορε διατάξει μέσω των διαφόρων αποφάσεων, διδοχικών αποφάσεων σύνδεση που είχαμε και τι προβλέπεται για την περίοδο μετά το 2020. Θέλουμε εδώ πέρα κάποιε διευκρινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το προτινόμενο χρηματοοικονομικό μέσο. Σύμφωνα με το 11ο ε, EDF προβλεπόντουσαν 5 εκατομμύρια, τα οποία δεν φαίνονται με απόλυτη σαφήνεια στη νέα αυτή προτινόμενη απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλαμε να γνωρίσουμε λοιπόν αν μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας προβλέπονται κάποια νέα ποσά και αν μπορούμε να κρατήσουμε επίσης και το απόθεμα εκείνο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την επανοικοδόμηση μετά από φυσικές καταστροφές. Επίσης θέλαμε να γνωρίζουμε αν υπάρχει μία συνέργεια μεταξύ των δραστηριοτήτων επίγουσας δράσης, καθώς επίσης και των αποθεμάτων που προβλέπονται στο δικό μας το χρηματοδοτικό κονδύλιο. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να κρατήσουμε το υφιστάμενο αυτό απόθεμα. Πρέπει να δούμε, αν δεν διατηρηθεί το απόθεμα αυτό, πώς θα χρηματοδοτηθούν οι δράσεις ανοικοδόμησης μετά από φυσικές καταστροφές ή αν προβλέπεται μείωση για αυτές τις δράσεις. Πιστεύουμε ότι μόνο αύξηση θα πρέπει να δούμε, γιατί ιδίω μετά το 2017 υπήρχαν πάρα πολλά υπερπόντια, δάφοι εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετώπισαν πολλές φυσικές καταστροφές, ιδίω μέσω καταιγίδων ε, η ίδια η Γρελανδία πλήγει από τσουνάμι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να χρηματοδοτεί όλες αυτές τις προσπάθειες ανοικοδόμησης μετά τις ε, φυσικές καταστροφές. Οι κανόνες που έχουν να κάνουν με την χρηματοοικονομική υποστήριξη. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια νέα ευελιξία η πολιτή αυτή αρχή νέα η οποία προβλέπεται, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία για μας και επίση δεν είναι σαφές αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα κονδύλια εκείνα τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή αν αυτά τελικά ακυρώνονται. Χρειαζόμαστε επίση πιο απλουστευμένου κανόνε για τον προγραμματισμό που επιτελούν τα υπερπόντια εδάφη. Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία τα υπερπόντια εδάφη και υπερπόντιες χώρες έχουν ζητήσει ε, πιο ευέλικτους μηχανισμούς οι οποίοι θα μπορούσαν να προωθήσουν ε, όχι μόνο τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την ε, περιφερειακή συνεργασία με άλλες όμορες περιφέρειες και χώρες. Θα θέλαμε περισσότερες διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς μπορεί αυτή η προσέγγιση να εφαρμοστεί στην πράξη. Επίσης είναι σημαντικό να μπορούν να συμμετέχουν τα υπερπόντια εδάφη και στον προγραμματισμό και την επιλεξιμότητα προγραμμάτων στα πλαίσια του DCI. Θα θέλαμε λοιπόν ως ηχέα να είμαστε επιλέξιμα για τα θεματικά αυτά προγράμματα. Από την άλλη όμως τονίσουμε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε προκειμένου να υποφεληθούμε από τα προγράμματα αυτά. Για παράδειγμα, έχουμε ελάχιστε επενδύσεις αυτή τη στιγμή σε υπερπόντιες χώρες και δάφη στα πλαίσια του DCI. Τώρα, όσον αφορά τα ενωσιακά προγράμματα, είμαστε ικανοποιημένοι με τις βασικέ βασικές αρχές οι οποίες έχουν διατηρηθεί στη νέα απόφαση για σύνδεση των ΙΧΕ. Η προσβασιμότητα όμω αποτελεί πρόκληση από το 2014 στο 2018, 125 προγράμματα, εκ των οποίων 65 ήταν οι υποφελούμενοι από τις ΙΧΕ. 6 εκατομμύρια περίπου δόθηκαν και δύο εκ των τριών προγραμμάτων είχαν να κάνουν με το Erasmus Plus. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να προβλεφθούν περισσότερα μέτρα υπέρ των ΙΧΕ και στο νέο άρθρο το προ 94 μάλλον του ΟΑΔ, της απόφασης για τη σύνδεση των ΙΧΕ, θα πρέπει να προβλέπονται νέες διατάξεις που να διευκολύνουν την επιλεξιμότητα και την πρόσβαση των ΙΧΕ. Στα πλαίσια του 94.3, του άρθρου 94.3 προβλέπεται ότι θα πρέπει οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη να υποβάλουν αναφορές για τη συμμετοχή τους σε νοσιακά προγράμματα. Στο άρθρο 83.3 προβλέπεται ότι θα πρέπει να υποβάλουμε εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την συμμετοχή μας σε νοσιακά προγράμματα κάθε χρόνο από το 2020 και μετά. Η ΟΚΤΑ συλλέγει τα τελευταία χρόνια δεδομένα και πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχει αλληλοπικάλυψη των προσπαθειών. Επίσης θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι οι αρμόδιες δυτικές αρχές δεν ενημερώνονται πάντα για τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν οι ΙΧΕ και το θέμα είναι ότι δεν έχει ζητηθεί στο παρελθόν από υπερπόντιες περιφέρειες να εκπονούν τέτοιες εκθέσεις. Επίσης, το ποσό το οποίο προβλέπεται ω χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή για τη ΣΥΧΕ δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση να υπομισθούν την αρμοδιότητα αυτή οι βρεπόντιε χώρε και εδάφη. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να εκπονεί αυτέ τι εκθέσει. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ, Κάρολ. Όπω είπα, συγγήτρια δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ. Ο συγγητή δεν μπορεί να παραβρεθεί. Όμως, θα δώσουμε τώρα το λόγο στην Συριάννα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να παρουσιάσω την θέση της, ε, του εισηγητή για της ε, είχε βρίσκεται στη Νέα Καλλιδονία για λόγους υγείας και μου ζήτησε να σας ε, ζητήσω συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και να παρουσιάσω τη θέση του. Καταρχήν ο κύριος Πόγκα θέλει να ευχαριστήσει την Επιτροπή για την εξαιρετική ε, πρότασή της, η οποία αντιστοιχεί στην θέση του Κοινοβουλίου για τις είχε, δηλαδή να υπάρχει ένα μοναδικό και ειδικό εργαλείο για τις είχε αυτό το OED ισχύει για όλες τις είχε, περιλαμβανομένης της, Ιρλαν... της Γρυλανδίας και παρέχει βοήθεια σε αυτή την εταιρική σχέση. Οπότε υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα, απλουστεύεται ο μηχανισμός και υπάρχει διαφάνεια και εξουσίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά το περιεχόμενο του OED, ο κύριος Πόγκα θέλει να πει τα εξής πέντε. Πρώτον, τα νέα OED ε θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, του SDG και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, πρόθεση της ε, ισότητας ανδρών και γυναικών που περιλαμβάνονται στις συνθήκες. Δεύτερον, η περιφερειακή ε, ολοκλήρωση των είχε θα πρέπει να συμπεριληφθεί ε, στον ενισχυμένο διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει στις είχε καθεστώς παρατηρητή στις, στις επαφές με τις τρίτες χώρες αφενός και κατά τρίτον και κατά δεύτερον τέτοιες χώρες θα πρέπει να προσκαλούνται στα πιο πολιτικ... στο πιο πολιτικό φόρουμ ή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι πολιτικές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις απόψεις και τις δυσκολίες των είχε. Η είχε ε, ε, είναι κομμάτι των... της ευρωπαϊκής οικογένειας και άρα είναι επιλέξιμα για τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αναφέρει το άρθρο 83 του ODA. Ο κύριος Πόγκα θεωρεί ότι ε, ε, το Συμβούλιο του OED θα πρέπει να επιμείνει περισσότερο όσον αφορά την επιλεξιμότητα των είχε στο Εράσμους και σε μια σειρά από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις, ε, τα συμφέροντα των είχε όταν διαπραγματεύεται συμφωνίες ελευθέρων εμπορίου με τρίτες χώρες. Επιπλέον, όλα, όλος ο προγραμματισμός θα πρέπει να περιληφθεί στον OED. Ε Δεν έχει νόημα την, ε, η υλοποίηση ε, του, του προγραμματισμού NDICI, γιατί αυτό το οποίο περιλαμβάνεται τώρα στην τρέχουσα απόφαση για τη Γρυλανδία να ισχύσει για, τους υπόλοιπους, για τις είχε. Αυτό θα μπορεί να γίνει ένα μέσον για για τα είχε, για να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες του. ο χρηματοδοτικός φάκελος πρέπει να αυξηθεί στα 669 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχεί στο τρέχον επίπεδο χρηματοδότησης. Επιπλέον, ο επαναπατρισμός μεταξύ είχε πρέπει να είναι πιο, πιο ισορροπημένος. Η ένταση βοήθειας για κάθε είχε θα πρέπει να, να στηρίζεται σε διαφανή κριτήρια και να υπάρχει ένας εδαφικός φάκελος. Ο κύριο Πόγκα ε, θα παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης στις 20 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε τώρα να δώσουμε το λόγο στους υπόλοιπους και κοιόδης, συγητές και λοιπούς συναδέλφους. Ντόρου Φρουντζουλίκα είναι ο πρώτος. Πάρα πολύ ωραία το προφέρατε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Και τη κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι οι σχέσεις με τη ΣΥΧΕ και τη Γρυλανδία πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η πολιτικο-οικονομική και κοινωνική συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί μέσω αυτής της νέας συμφωνίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικέ σχέσεις, τις ιστορικούς δεσμούς και τις εταιρικέ σχέσεις που έχουμε με αυτές τις χώρες ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε μια θετική πρόθεση, να υπάρξει δηλαδή απλούστευση λόγω της, μέσω της συγχώνευσης, για να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα. Γιατί οι πολιτικές σχέσεις με ηχέ και η χρηματοοικονομική πρώτη πόρη θα τεθούν κάτω από το ίδιο εργαλείο. Και θα βοηθήσει και διοικητικά αυτό, θα δημιουργηθούν νέε συνέργειες, θα βοηθήσουν την καλύτερη εφαρμογή. Συμφωνούμε για το βασικό στόχο, σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Σύνδεσης. Τρεις είναι βασικοί πιλότες. μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, μεγαλύτερη αφεκτικότητα και λιγότερη, ε, λιγότερα τροτά σημεία. Είναι σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι η μελλοντική συνεργασία έχει ένωσης θα πρέπει για να εφαρμόσει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και τη συμφωνία του Παρισιού. Και ελπίζουμε οι δράσεις να βάζουν ε, την έμφαση στις διασυνδέσεις και στις ε, ολοκληρωμένες δράσεις για την επίτευξη πολλαπλών στόχων με συνεκτικό τρόπο. Τέλος, θέλω να προσθέσω δύο λόγια για την Γρυλανδία. Θεωρώ ότι είναι θετικό τα επιτεύγματα της απόφασης να μην χαθούν. Θα πρέπει να, δοθούν, ε, να δοθεί έμφαση στις ιδιαιτερότητες της σχέσης με τη Γρυλανδία. Σχέσεις ιστορικές μεταξύ Ένωσης, Δανίας και Γρυλανδίας πρέπει να διατηρηθούν, να διαφυλαχθούν. Έχουμε ένα έγγραφο για τη Συμφωνία της Γρυλανδίας με βασικό στόχο τη διατήρηση ακριβώς των μονοκρέων σχέσεων και πρόθεση της αεφόρο ανάπτυξη στην Ολλανδία. Αυτό μέχρι στιγμή το έχουμε πετύχει, πρέπει όμω να συνεχιστεί και μετά το 2020. Maria Hoibuch είναι η επόμενη μιλητέ. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να μιλήσω για τη σημασία που έχει συνεργασία σε ό,τι αφορά ε, τα ε, υπερπόντια εδάφη και χώρες. Ε, υπόθηκαν πολλά και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Έχω κάποιες ερωτήσεις για κάποια σημεία που θέλω να σχολιάσω. Το πρώτο, η πρόταση μιλά για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στην Ανατολική Σκέψη 9 λέει ότι στο πλαίσιο αυτή τη απόφαση θα πρέπει να, ελαφο... να υιοθετηθούν ε, μέτρα για την ε, επίτευξη αυτών των στόχων ε, και να δώσουμε επίσης έμφαση στην συνεκτικότητα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτούς τους στόχους. Ωραία είναι αυτά. Όμως δεν υπάρχουν λεπτομέρειες μετά στο κείμενο ως προς αυτό για τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε, για τη βιωσιμότητα για παράδειγμα. Γιατί λέτε εδώ για μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν, αλλά δεν βλέπουμε κάτι συγκεκριμένο και ότι πρέπει να υπάρχει προσαρμογή αυτών που εφαρμόζονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Για το μέλλον τώρα. Σε αυτά τα είχε. Υπάρχει περιορισμένο ανθρωπικό δυναμικό και μέσα διοικητικά και πόροι. Και δεν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν οι στόχοι του προγράμματος. Στην ετολογική σκέψη το αναφέρουμε, αλλά δεν είναι σαφές στην πράξη πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ώστε να μπορούν τα κράτη να εφαρμόσουν και να αξιοποιήσουν αυτά τα προγράμματα καλύτερα. Και επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, ε, σε ό,τι αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, συνολικά ο στόχος της Κομισιόν είναι το 25% των δαπανών της Ένωσης ε, να ε, υπηρετεί ε, τους στόχους για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτού έχουμε 20% μόνο για το κλίμα. Γιατί. Γιατί είναι χαμηλότερο το ποσοστό εδώ σε σχέση με αυτό το οποίο έχει αποφασίσει συνολικά η Ένωση. Και τέλος, μια παρατήρηση για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ευέλικτοι, όπως προβλέπετε σε αυτή την πρόταση, ε, πρέπει να προωθήσουμε τα μέτρα τα οποία απαιτούνται. Ευχαριστώ πολύ ήταν οι ερωτήσεις, Μαρία. Ελπίζω αργότερα να έχουμε και απαντήσεις. Τελευταίος, ο κύριος Τσέλερ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αυτά τα νησιά, αυτά τα εδάφη που είναι κατάλοιπα της απεικιοκρατικής εποχής, τέλος πάντων, δεν θέλουν να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε όσα τις εξόχους από κέντρες περιφέρειες, όπου ισχύουν οι νόμοι και οι διάφοροι άλλοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το δυναμικό και από την άλλη πλευρά, όταν χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια, πρέπει να μπορεί να παρέχεται αυτή. Στο πλαίσιο τώρα της αναπτυξιακής συνεργασίας το πρόβλημα που προκύπτει με αυτά τα νησιωτικά κράτη, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι νησιωτικά κράτη, έχει να κάνει και με μια συζήτηση που γίνεται σε ό,τι αφορά την ε, ε, φορολόγηση. Δεν πληρώνουν πολλοί ε, φόρους, ε, υπάρχουν φορολογική παράδειση εκεί και υπάρχει αυτό λίγο, δημιουργεί κάποιες αντιφάσεις. Δηλαδή θέλουν βοήθεια από τη μία, αλλά από την άλλη πλευρά παρέχουν φορολογικούς παραδείσους για αυτούς που δεν θέλουν να πληρώσουν φόρους. Πρέπει να το δούμε νομίζω και αυτό στη συζήτηση που έχουμε. Είχαμε τα Paradise Papers, τα Panama Papers. Νομίζω ότι το θέμα εδώ είναι η διαφάνεια. Θέλουμε να υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ζητήσουμε και από τις χώρες αυτές με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε και τις απαντήσεις τώρα Ενδεχομένως πρώτα η κυρία Μιλό. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τι ερωτήσει αυτέ και για τι παρατηρήσει που κάνατε, που θεωρώ ότι εν γέννη είναι θετικέ και ουσιαστικά φαίνεται να αξιολογούν θετικά τι αλλαγέ που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση σύνδεση. Αυτό φάνηκε από τι διάφορε παρεμβάσει. Τώρα, πιο συγκεκριμένο. όσον αφορά τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Υπάρχουν ορισμένες οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν, που έχουν να κάνουν βασικά με τον στόχο, τους στόχους που πρέπει να πετύχουν οι ΙΧΕ, η πρόθεση της ισότητας των φύλων μεταξύ άλλων. Πιστεύω προφανώς ότι όλες οι δράσεις συνεργασίας και όλοι οι τομείς συνεργασίας που απαριθμούνται στην απόφαση αυτή ανταποκρίνονται σε ένα πεδίο δράσης το οποίο είναι ιδιαίτερα ευρύ, αλλά μπορούν να οι αυτές να ομαδοποιηθούν, να συντονιστούν μεταξύ τους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Ξέρετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η διατύπωση που χρησιμοποιούμε και στις διαπραγματεύσει που θα λάβουν χώρα με τα κράτη-μέλη. Πάντως νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο στόχος της εν λόγω συνεργασίας είναι να πετύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Το ίδιο και το στόχο της ισότητας των φύλων. Και αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται στη διατύπωση που χρησιμοποιούμε. Όσον αφορά τώρα το ποσό, καθώς επίσης και την υλοποίηση τελικά της συνεργασίας. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλά πράγματα θεσπίζονται. Για παράδειγμα, πώς θα χρησιμοποιηθούν τα υπόλοιπα μέσα συνεργασίας, τι θα γίνει με το μελλοντικό προπολογισμό, τι θα γίνει με το μηχανισμό υλοποίησης. Όλα αυτά βρίσκονται υπό συζήτηση στις διάφορες αρμόδιες ομάδες, άρα είναι πολύ νωρί αυτή τη στιγμή να πούμε επίση με απόλυτη σαφήνεια πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά στην πράξη. Ωστόσο, η πιο σημαντική ανησυχία που ακολουθείται πιο συχνά, που αναφέρεται, με συγχωρείτε, πιο συχνά, είναι ότι οι υπερπόντιες χώρες και τα υπερπόντια εδάφη δεν καταφέρουν να υποφεληθούν στην πράξη από αυτή τη συνεργασία. Εμείς επιβεβαιώνουμε πραγματικά τη βούληση αλλά και τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρχει ένας ελαφρύς, αν θέλετε, προγραμματισμός για τη Συχέ. Αυτό προτείνεται και στην πρόταση απόφαση. αυτό κάνουμε μέχρι στιγμή και ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό ακριβώ θέλουμε να προωθήσουμε και αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση στου επόμενου μήνε, προκειμένου να βρεθούν συγκεκριμένοι μέθοδοι συνεργασία για να μπορέσουν να αποφεληθούν από τα συγκεκριμένα κονδύλια που προβλέπονται για τα εδάφια αυτά οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι. Επίση, ενδεχομένω θα πρέπει να χρησιμοποιούμε καλύτερα τα εφιστάμενα κονδύλια προκειμένου να στηρίξουμε τη ΙΧΕ και να καταφέρουμε να αποφεληθούμε από έναν πιο αποτελεσματικό προγραμματισμό και να καταφέρουμε να αποφεληθούμε από τα οριζόντια προγράμματα συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρόπο πιο έντονο. Νομίζω λοιπόν ότι σαφώς θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την τεχνική αυτή πτυχή της συνεργασίας. Όσον αφορά τώρα τον πολιτικό διάλογο, Νομίζω ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους και ένα από τα βασικά στοιχεία που βλέπουμε στην απόφαση αυτή, στο σχέδιο απόφασης. Ο πολιτικός διάλογος διεκπεραιώνεται μέσω των συγκεκριμένων διάβλων που προβλέπονται στην απόφαση αυτή. Μπορεί ο διάλογος να είναι διμερής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών μελών και ΙΧΕ και προφανώς είμαστε απόλυτα διαλλακτικοί και ενθαρρύνουμε κιόλας θα έλεγα έναν ενισχυμένο πολιτικό διάλογο. continue or yeah, je cherchais quelque chose. Okay. euh... Ok, ce sera bon. Euh... Well, I can um, reference. Uh... Λοιπόν, μπορώ να αναφερθώ στην ερώτηση της κυρίας Σέλλερ για τους φορολογικούς παραδείσους κατάλαβα ότι έχουν αναλυφθεί δεσμέσεις για να γίνουν αλλαγές μέχρι το τέλος του 2018 και έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις μεταξύ των, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της, των συγκεκριμένων υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, για τη συζήτηση αυτή η οποία μας έδωσε πολλές ιδέες για να προχωρήσουμε, αλλά και απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε τώρα στη συνέχεια. We continue to... Συνεχίζουμε με το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Επιτροπή μας συχνά συντάσσει γνωμοδοτήσεις επί των ε, αλληλευτικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναπτυσσόμενες χώρες για τον λόγο ότι η, τα ψάρια είναι μια, ε, μια πολύτιμη πηγή ε, πιστιστικής ασφάλειας, θέσεων εργασίας και ανάπτυξης. Η δυνατότητα των αναπτυσσομένων χωρών να υποφεληθούν από τους ληφτικούς τους σπόρους και μάλιστα με βιώσιμο τρόπο πρέπει να προστατευτεί και να ενισχυθεί. Η βιώσιμη αλία είναι κομμάτι αυτού που χρειάζεται για την προστασία και την βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλασσίων πόρων. Πρόκειται για τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης συμπαριθμών 14. Τώρα θα δούμε πιο προσεκτικά αυτόν τον συγκεκριμένο στόχο ε, βιώσιμης ανάπτυξης και τους στόχους που ε, τον αφορούν με ε, έμφαση στο τι διακυβεύεται για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ε, το στόχο αυτό με διάφορους τρόπους. Επηρεάζει το Ελληνίνιο και άλλα θαλάσσια ρεύματα, ανεβάζει το επίπεδο των θαλασσών και αλλοιώνει τα οικοσυστήματα των ε, αλλιευτικών αποθεμάτων που χρησιμοποιούνται με την πρόκληση απολειών και ανάγκης προσαρμογής. Οι ιδέες για την διεύρυνση της γαλάζιας οικονομίας χρειάζεται να μελετηθούν προσεκτικά. Ε, τι υπόσχονται αυτές οι ιδέες για, την, ε, για τις αναπτυσσόμενες χώρες και ποιους κινδύνους για να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε το πώς, αντιλαμ... το πώς αντιλαμβανόμαστε τα θέματα αυτά, έχουμε προσκαλέσει τον επικεφαλής του προγράμματος ε, ΟΗΕ ε, στις Βρυξέλλες, τον κύριο Τιερή Λούκας. Σας ευχαριστώ κύριε Λούκας που ε, συμφωνήσατε να μας κάνετε μια εισαγωγή περίπου 7-8 λεπτών επί του θέματος. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης. Θα ε, αναφερθώ στον ε, στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 14 και τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, ο, η επικεφαλής, ο επικεφαλής οργανισμός του ΟΗΕ για την ε, κλιματική αλλαγή έχει θέσει ένα θεματολόγιο και ε, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες για το παγκόσμιο περιβάλλον. Έχουμε ε, ασχοληθεί ε, με το θέμα αυτό του στόχου υπαριθμών 14 στο, σχετικά με το στόχο 14 υπάρχουν 10 δείκτες. Λόγω του περιορισμένου χρόνου δεν θα αναφερθώ σε όλους, αλλά θα αναφερθώ μόνο στους 5 πρώτους. Πρώτον, την θαλάσσια ρήπανση και αυτό είναι σημαντικό γιατί ε, το περιβάλλον... Ε, ε, ο οργανισμός μας και με τον κύριο Τίμεμανς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την ρήπανση των, με πλαστικά που είναι σημαντικά για τα νησιά. Επίσης, ο δεύτερος δείκτης, γιατί είναι σημαντικό να ε, ε, γίνεται βιώσιμος χειρισμός της αλίας. Μια δουλειά που εμείς ως άνθρωποι, εμείς οι, άνθρωποι που κατοικούν στη στεριά δεν το προσέχουμε αρκετά και υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία που είπατε για τη γαλάζια οικονομία. Θα αναφερθώ επίσης στους δείκτες 3, 4 και 5 πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αύξηση της οξύτητας των ωκεανών που είναι απειλή για ε, τους ε, ωκεανούς. Ε, αυτό επηρεάζει, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και τις, τους υφάλους, τους καρολογενείς υφάλους που είναι φυτόρια, είναι όπου γεννιούνται τα ψάρια. Και επίσης θα αναφερθώ στον δείκτη 5, το τι μπορείτε να κάνετε δηλαδή για να προστατευτεί το 10% των ε, παράκτιων και θαλασσίων περιοχών και το 6% και θα γίνει ε, μια σημαντική σχετική συνάντηση στο τέλος χρονιάς. Άρα, από σήμερα η παγκόσμια τάση και παίρνω τα στοιχεία από το ε, πιο πρόσφατο πολιτικό φόρουμ υψηλού επίπεδου και ε, την έκθεσή μας για το παγκόσμιο ε, ε, περιβάλλον. Το 40% των παγκοσμίων των ωκεανών του κόσμου επηρεάζονται σημαντικά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, περιλαμβανομένες και της ρήπανσης. Και δεύτερο, οι επιδοτήσεις για την αλία, και θα εξηγήσω τι είναι επιδοτήσεις, οι αρνητικές επιδοτήσεις έχουν αρνητικό αποτέλεσμα και έχει υπολογιστεί ότι χάνουμε περίπου 50 δις κάθε χρόνο λόγω αυτών των ε, κακών επιδοτήσεων. Δεν γίνεται διαχείριση αλίας με τρόπο βιώσιμο. Επίσης, όπως είπα, σημαντικό είναι να γνωρίσουμε ότι το 20% των θαλασσίων οικοσυστημάτων θα πληγούν από την μόλυνση και την ε, νητροποίηση με βάση τους υπολογισμούς. Και αυτό θα επηρεάσει το, ε, τον ευτροφισμό μέχρι το 2050. Επίσης, κάποια στοιχεία τα αποθέματα ψαριών. Ήταν το 74-90%, τώρα είναι στο 69% ακόμα. Δεν είναι τόσο κακό ακόμα. Θα δείτε όμως ότι πολλά από τα μεγάλα ψάρια στα οποία επενδύουμε πολύ έχουν ε, επηρεαστεί και αυτό επηρεάζει πολλές χώρες. Η οξύτητα της θάλασσας έχει αυξηθεί κατά 26% και αυτό επηρεάζεται από την ε, κλιματική αλλαγή και πρέπει να αλλάξει. Έχουμε και κάποιες θετικές τάσεις σε θέματα που αφορούν τη θάλασσα. 16% ε, των θαλασσίων υδάτων τώρα προστατεύονται και αυτά λόγω της εθνικής δικαιοδοσίας και, και έχουμε από, αλλαγή από το 30% στο 44% τους ε, κρίσιμους ε, θαλάσσιους χώρους βιοποικιλότητας. Κάποιες τάσεις, αν δείτε τα νούμερα από τη δεκαετία του 50 για την επιτρεπόμενη έκταση της βιομηχανικής αλίας στην Αναπτυξιακή Επιτροπή, όταν αναφερόμαστε στις χώρες Αφρική Αφρικής, μιλάμε για το δεύτερο σχεδιάγραμμα και βλέπουμε ότι έχουμε μια αύξηση από 10 σε 20 εκατομμύρια σε 60 χρόνια, ενώ πήγαμε από 50 σε 80 σε το βιομηχανικό επίπεδο. Και αυτό είναι θέμα, διότι το μερίδιο των θαλασσίων πόρων δεν κατανέμεται εξίσου ανάμεσα στις χώρες και στο επόμενο σχεδιάγραμμα θα το εξηγήσω αυτό. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Αυτό που έχει σημασία είναι εδώ να διαπιστώσουμε ότι ποια είναι η κατανάλωση των ψαριών και των ε, θαλασσινών σε σχέση με το ΑΕΠ. Το χαμηλότερο το ΑΕΠ, ε, τόσο ψηλότερο η ε, κατανάλωση. Η, Καμ, η Καμπόζη, η Γκάμπια, και η Χρυπάτη και η Γκάνα, οι χώρες αυτές είναι αυτές που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, να επηρεαστούν, γιατί το 17% του παγκόσμιου πληθυσμού ε, προσλαμβάνει τροφές από την, από την αλία, αλλά στις χώρες αυτές το ποσοστό είναι ψηλότερο. Κάτι άλλο σημαντικό είναι η τάση της ηχθειοκαλλιέργειας και της ε, ε, τι, αυτό αυξάνει, αλλά τι μπορεί να γίνει για να αυξηθεί αυτό και στην Αφρική και μάλιστα με τρόπο βιώσιμο και κάποια θετικά μηνύματα. Αυτό που έχει προβληθεί είναι η νέα βιώσιμη πιστοποίηση τροφών, ε, δηλαδή τα Marine ε, Stewardship Council, ε, το Aquaculture Stewardship Certification κλπ. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κομμάτι της γαλάζιας οικονομίας για την παραγωγή τροφών και πρωτεϊνών για ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίως λόγω, μέσα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Εν κατακλείδη, το, γίνεται μεγάλες διαπραγματεύσεις στο Buenos Aires στο πλαίσιο του ΠΟΕ, για, που είναι ευκαιρία για να σταματήσουν οι επιδοτήσεις της αλίας Σαφώς οι χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να επιδοτούν τα καύσιμα, τα μεγαλύτερα σκάφη κλπ. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι η λύση για το μέλλον της αλίας. Είναι κάτι που πρέπει όλοι να το αντιληφθούμε. Και ο δείκτης υπαρθμών 6 είναι επίσης σημαντικός. Και τέλος θα κλείσω με την ε, ε, εκστρατεία του περιβάλλοντος του ΟΗΕ για τις καθαρές θάλασσες είναι σημαντικό για όλους να έχουμε καθαρές θάλασσες ή, ή, μόλις με πλαστικά επηρεάζει τις θάλασσες κυρίως τις χώρες χαμηλού εισοδήματος επηρεάζει όμως και την τροφική αλυσίδα και αυτό το μετράμε τώρα. Πώς μπαίνει το πλαστικό στα ψάρια και από εκεί μέσω αυτών στο σώμα μας και αυτό είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί για λόγους υγείας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή Many thanks. It's, it's a great pleasure to, to hear this presentation. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Οι βουλευτές, θέλετε το λόγο παρακαλώ. Έχετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις για κάτι, οτιδήποτε. Όχι. Να, Μαρία. Yeah, Μήπως να βάλετε και ακουστικά. Δεν είμαι και η ε, στα θέματα της αλίας, ε, αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό το γράφημα που δείξατε με τις διάφορες ε, αληφτικές μεθόδους που δείξατε σε σχέση ιδίως με τη βιομηχανική αλία που έχει σημειώσει μεγάλη άνοδο. Είναι παραδοσιακή αλικία, πολύ λίγη ανωδική τάση παρουσιάζει θα μπορούσατε να μας πείτε σε ό,τι αφορά τις αληφτικές συμφωνίες και την αληφτική νομοθεσία, τι μπορεί να κάνει για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και να παρεμποδίσουμε αυτή την τάση κατά κάποιο τρόπο και να μπορέσουμε εκεί που υπάρχει παραδοσιακή αλία να βοηθήσουμε δεν ξέρω, και ίσως μπορούμε να πάρουμε και τα ε, μεγάλα σκάφη από τις θάλασσες. Ε, πόση αλληλευτική δραστηριότητα αντέχει η θάλασσά μας. Ε, αυτό περίπου θέλω να μάθω. Πρόεδρος, θα έπρεπε ίσως να αναφέρω ότι είμαι κόρη ψαρά εγώ και όλη η οικογένειά μου ζει από την Αλία. και είδα τα τελευταία 20-30 χρόνια ότι κάτι γίνεται με το νερό, ζεσταίνεται το νερό. Τα ψάρια είναι πολλά μένα, αλλά είναι άλλα είδη από αυτά που είχαμε εμείς. Και όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Και πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται στους ωκεανούς μας και τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να εξακολουθήσουμε να έχουμε από θέματα αλλήλων, μάλλον ε, ψαριών και αλληλευτική δραστηριότητα. Κύριος Τσέλερ, ευχαριστώ και θέλω να σας ευχαριστήσω για τα εντυπωσιακά νούμερα που μας είπατε, ε, που μας δείξετε. Δύο πράγματα μου χτύπησαν. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες ε, τις αλληλευτικές που βρέθηκαν εκεί διάφορα ε, στοιχεία, κάποια κενά ε, και σε σχέση με τις πληρωμές που δίνονται για τον Ευρωπαϊκό Ελευτικό Στόλο που κατά το 80% αποτελείται από μεγάλα ισπανικά σκάφη, κλείνει παρένθεση, ε, και τι γίνεται στα χωρικά ύδατα που μπορούν να ψαρεύουν και στις ακτές της ε, Βόρειας Αφρικής. Και το πλεόνασμα ήταν το δεύτερο, το surplus, σε ό,τι αφορά τα αποθέματα. Πώς μπορούμε ε, να ε, περιορίσουμε κάπως το, την αλληλευτική δραστηριότητα για να χαλαρώσει κάπως η κατάσταση. Υπάρχει αυτό το πλεόνασμα. Απ' την άλλη λέτε χρειάζεται επιστημονική παρακολούθηση, επιτήρηση. Στα εθνικά χωρικά υδατά, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται αυτό, ιδίως στα ψώμενα κράτη και απ' την άλλη πλευρά ο μεγάλος αλληλευτικός στόλος ε, που δραστηριοποιείται στα διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά, δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Σε ό,τι αφορά πάντα τις αλευτικές συμφωνίες, μας δείξατε κάποια νούμερα, κάποια ποσά. Για πλεονάσματα μας είπατε, αλλά μετά μας είπατε ότι συμφωνούμε κάποιες αλληλευτικές ποσοστώσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν επιτευχθεί, δεν φτάνουν σε, αυτό, σε αυτές τις ποσοστώσεις. Φτάνουν τα περισσότερα αυτά ε, αλλιεύματα στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Δεν ξέρω μήπως ε, κάποια κράτη πληρώνουν καλύτερα τα ορισμένα είδη ψαριών από ό,τι ίσως κάποια άλλα ε, ευρωπαϊκά κράτη. Αν δεν κάνεις για το στο για παράδειγμα. Φτάνουν εκεί ε, πολλά ψάρια από ευρωπαϊκό αλληλευτικό στόλο, γιατί επιτυχάνουν καλύτερη τιμή ψαράδες. Δεν πάνε και όλα τέλεια δηλαδή. Αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους, αν θέλουμε και η επόμενη γενιά ε, να μπορεί να βάζει σκάφη στις θάλασσες, ε, τι πρέπει να κάνουμε, ποιες είναι οι προτάσεις σας. Thank you very much. Then we have... Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι από την DG Mare. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. που Προσπαθήσατε να προφέρετε το επίθετό μου, το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε το λόγο σε εμά που εκπροσωπούμε την DG Mare της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακολουθήσαμε την παρουσίαση του κυρίου Λούκας, τον οποίο ευχαριστούμε και για τη σφαιρική αυτή παρουσίαση που έκανε όσον αφορά τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης παριθμών 14. Αυτός είναι και ο δικός μας ο στόχος στη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ. Η υγιής ωκεανή είναι πάρα πολύ σημαντική και για τη δική μας τη ζωή και γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχουμε και αυτόν τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης του υπαριθμό 14. Οι ωκεανοί αποτελούν σημαντική πηγή τροφίμων, εσόδων για ένα μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζουν πάρα πολύ το κλίμα, παρέχουν οξυγόνο στον πλανήτη μας και γι' αυτό ακριβώς το λόγο χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν το 2015 τα Ηνωμένα Έθνη αποφάσισαν να καταρτήσουν αυτούς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και θεώρησαν ότι ένας στόχος θα πρέπει να αφορά ακριβώς τους ωκεανούς, ο στόχος παριθμών 14. Δυστυχώς όμως οι ωκεανοί, όπως τα ακούσατε, υφίστανται πάρα πολλές πιέσεις, όπως η μόλυνση, η ρήπανση, η εξόριξη πόρων, η παράνομη αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλία, οι κλιματικές αλλαγές και η υπεραλίευση. Βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στους ωκεανούς και θα έλεγα ότι το τελευταίο έτος ήταν πραγματικά ένα έτος αφιερωμένο στους με μια σημαντική συνεδρία στον Ιούνιο στα Ηνωμένα Έθνη όπου στόχος συνεδρίασης αυτής ήταν ε, η μέθοδη επίτευξης του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 και τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε μια δική της συνδιάσκεψη με στόχο μάλλον με θέμα ότι η ωκεανοί είναι το μέλλον μας, όπου είχαμε εδώ πέρα πάρα πολλούς συμμετέχοντες από τον δημόσιο και το ειδικό τομέα, πάρα πολύ εμπλεκόμενοι στην προστασία των ωκεανών. Θα ήθελα πολύ γρήγορα να σας παρουσιάσω τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη του στόχου 14. Όλες οι θαλάσσιες πολιτικές αλλά και παράκτιες πολιτικές που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν ένα πλαίσιο για μια σφαιρική προσέγγιση της διαχείρισης των ωκεανών. Το θεματολόγιο το οποίο εγκρίναμε το 2016 για τους ωκεανούς προβλέπει ένα γενικότερο πλαίσιο για την ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης των ωκεανών έτσι ώστε οι ωκεανοί να είναι ασφαλείς, καθαροί και να μπορούν να χρησιμοποιούνται και να τυχάουν μια εκμετάλλευση η οποία θα είναι, η οποία θα είναι ασφαλής και νόμιμη. Τρει είναι οι βασικέ προτεραιότητε αυτού του θεματολογίου. Πρώτον, θα πρέπει να ενισχύσουμε το παγκόσμιο πλαίσιο διακυβέρνηση των ωκεανών, να συμπληρωθούν δηλαδή τα εφιστάμενα κενά. Δεύτερον, θα πρέπει να μειωθεί η πίεση που ασκεί ωκεανού και να δημιουργηθούν οι συνθήκε για μία μπλε οικονομία και θα πρέπει να αυξήσουμε επίση την επιστημονική γνώση. αυτή είναι η τρίτη προτεραιότητα, επιστημονική γνώση για του ωκεανού. Έχουν καταβληθεί προσπάθειε και για τι τρει προτεραιότητε. Όσον αφορά την βελτίωση τη διεθνού διακυβέρνηση για του ωκεανού, επετεύχθη πρόοδο στα Ηνωμένα Έθνη, προκειμένου να έχουμε ένα νομικά δεσμευτικό όργανο στα πλαίσια τη Σύμβαση των Εθνών για το Θαλάσσιο Δίκαιο, το οποίο θα έχει να κάνει με την συντήρηση καθώς επίσης και με την βιώσιμη διαχείριση του θαλασσίου περιβάλλοντος, ιδίως και των περιοχών εκείνων που βρίσκονται εκτός συγκεκριμένης ε, ε, δικαιοδοσίας, νομικής δικαιοδοσίας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήδη την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η πρώτη συνεδρίαση για το νέο αυτό μέσο, το οποίο μάλιστα γνώρι, η οποία συνεδρίαση γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να αποφύγουμε στον Αρκτικό ωκεανό κάθε μορφή παράνομης και αδήλωτης αλίας. Εδώ πέρα υπάρχει μια συμφωνία την οποία πρόκειται να προσυπογράψουν πολλές χώρες. Επίσης, σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί και για τη μείωση της μόλυνσης. Έχουμε μια στρατηγική για τη μείωση πλαστικού και τη μείωση της μόλυνσης από το πλαστικό στις θάλασσες και στους ωκεανούς, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε πραγματικά να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή για την πρωτοβουλία αυτή, η οποία εντάσσεται στη γενικότερη ε, προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας. Επίσης, 23 κράτη-μέλη ενέλαβαν δράση για να εφαρμόσουν ε, την ε, οδηγία πλαίσιο για την στρατηγική για τις θάλασσες, ώστε να υπάρχει ένα καλύτερο καθεστώς και μια καλύτερη ποιότητα των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, Επίσης, έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε πάρα πολύ σημαντικά από τα 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχουμε επιπλέον 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα των προστατευομένων από το πρόγραμμα Natura ακτών και περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε μέσω πρωτοβουλειών όπως το BioPharma 2 με 22 εκατομμύρια ευρώ μάλιστα χρηματοδοτεί το πρόγραμμα αυτό με 7 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται, μάλλον υλοποιούνται άλλα προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με συνεργασία με τρίτε χώρε. Αυτά είναι λίγα από τα προγράμματα μόνο τα οποία θα μπορούσα να αναφέρω. Η συνάδελφο από την DG DEFCO μπορεί να σα μιλήσει περισσότερο για τα προγράμματα αυτά διεθνού συνεργασία, τα οποία προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την αλληλεία, και εδώ πέρα έχει επιτευχθεί πρόοδο μέσω τη έγκριση ενό νέου κανονισμού για την βιώσιμη εκμετάλλευση των εξωτερικών ε, στο, στόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία πρόταση που έχει γίνει επίση για την τροποποίηση του υφιστάμενου συστήματο ελέγχου των ελευτικών στόλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει και αυτή έτσι ώστε μέχρι το 2020 να καταργηθούν στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου συγκεκριμένε μορφέ ελευτικών επιδοτήσεων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να τηρήσουμε την καταληκτική ημερομηνία του 2020 που έχει τεθεί από τον στόχο βιώσιμη ανάπτυξη παριθμών 14. Επίση, έχουμε διεθνή συνεργασία αλλά και διμερεί επαφέ με τρίτες χώρες προκειμένου να <clears throat> προβλέπονται συγκεκριμένες κανόνες όσον αφορά την καταβολή δασμών. Επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε και να εξυγχρονίσουμε το σύστημα καταμέτρησης και χαρτογράφησης ε, των αλληλευτικών αποθεμάτων, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται περισσότερο, να χρησιμοποιείται περισσότερο συστήματα πληροφορικής. Επίσης, ε, μέσω της ΠΕΣΚΑΟ, της ΕΚΟΦΗΣ και άλλων προγραμμάτων έχουμε προωθήσει τις ε, αλλιευτικές διοικητικές ικανότητες τρίτων χωρών οι οποίες συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια του προγράμματος ε, Ορίζοντα 2020 έχουν δοθεί 260 εκατομμύρια σε τήσια βάση για προγράμματα επιστημονικά και ερευνητικά όσον αφορά την ε, βελτίωση της ποιότητας των ωκεανών. Επίσης, ε, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών. Διακόπτη Πρόεδρος, πιέζει ο χρόνος. Αν μπορείτε, παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε. Ήθελα απλώς να σας πω ότι σε σχέση με την τα επόμενα στάδια, είναι σημαντικό να δούμε ότι στο πλαίσιο της, ε, διεθνού, της ανακοίνωσης για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών εκπονήσαμε μία μελέτη η οποία θα μας επιτρέψει να δούμε πώς μπορούμε να επεκτείνουμε τις ε, συμφωνίες ε, εταιρικής σχέσης για την αλία οι οποίες να περιλαμβάνουν πλέον και μία πτυχή η οποία θα έχει να κάνει με την ε, οικολογική βιώσιμη αλεία. Μπορούμε λοιπόν να δούμε πλέον στα πλαίσια των νέων αυτών ε, συμφωνιών πώ θα μπορούσαμε να εντάξουμε και την πτυχή που έχει να κάνει με το στόχο βιώσιμη ανάπτυξη παρελθόν 14. Επίση, η Eurostat ε, έχει πρόσφατα δημοσιεύσει την έκθεση πρόοδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και γίνεται και ειδική μνήα στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης παραθμό 14. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περάσουμε στις απαντήσεις. Οι σύντομες παρατηρήσεις, θέλει κανείς να κάνει κανένα σχόλιο, όχι. Απαντήσεις λοιπόν. Κάποιες απαντήσεις και περαιτέρω ανάγνωση ενδεχομένως. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Αυτό που είδαμε εμείς είναι μία έκρηξη της αλίας. Το είδαμε και στη Γεωργία όμως. Και ο τρόπος με τον οποίο συνολικά αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον ε, δημιούργησε θέματα. Αυτό που θέλω να σας πω για τις θάλασσες είναι ότι υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Και αν κάνουμε απλά πράγματα, θα δούμε αποτελέσματα μέσα σε 15-20 χρόνια. Όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Η καθηγήτρια ονομάζει τα σημεία αυτά σημεία ελπίδα και έχει εντοπίσει κάποια σημεία της γης όπου θα πρέπει να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον. Γιατί ξέρουμε ότι τα αποθέματα ε, ψαριών μπορούν να είναι σε χαμηλό επίπεδο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι κρίσιμα τα επίπεδα. Αλλά όταν υπάρχει νητροποίηση και μόλυνση, το πρόβλημα είναι σοβαρό. Έτσι λοιπόν, σημαντικό είναι ότι αν προστατευθούμε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον έντονο γεωγραφικό στοιχείο. Από σήμερα οι ε, εκθέσεις Οσεάνο 2011 Ισπανία ε, και άλλες δύο χώρες έχουν το μεγαλύτερο στόλο και άλλες μικρότερες μικρότερους τόλους. Πρέπει όμως οι χώρες αυτές να εφαρμόσουν τον κανονισμό. Πώς θα γίνει αυτό. Ο απλός τρόπος θα ήταν να γίνει μια συμφωνία με αυτές τις χώρες. Οποιαδήποτε χώρα, Σενεγάλη ή άλλες, η ακτή της Γουινέας. Μπορεί κανείς να γίνει μια συμφωνία παρόμοιες με αυτές που γίνονται για την βιώσιμη ανάπτυξη κάποιων τροφών. Να υπάρχει βιώσιμη χρήση των ψαριών. Η παρακολούθηση και η συμφωνία θα πρέπει να γίνεται από την κυβέρνηση. Να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εδώ βλέπω δύο πλεονεκτήματα. Πρώτον, ενισχύεται συνεργασία ε, Ευρω... Ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών. Θα δούνε τα ωφέλη και για την τοπική αλία αλλά και για την κυβέρνηση, γιατί τα χρήματα θα πάνε σε κυβερνητικό επίπεδο. Δεύτερον, θα δοθούν έντονες ενδείξεις στις μεγάλες χώρες που επηρεάζουν την περιοχή. Πολιτικά λοιπόν έχει νόημα αυτό. Και τέλος, γνωρίζουμε ότι οι χώρες αυτές θα δουν οικονομική ανάπτυξη και άρα μεγαλύτερη σταθερότητα. Εγώ αυτό θα έκανα. Φυσικά οι ενδείξεις βελτίωσης θα έρθουν γρήγορα, θα έχουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης και θα έχουμε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε τι γίνεται εκεί μια συμφωνία με τις χώρες αυτές ε, μπορεί να ενισχυθεί η δυνατότητά του σε εθνικό επίπεδο και δίνοντάς τη δυνατότητα να επιβάλλουν, να παρακολουθήσουν τις συμφωνίες αυτές, για μένα αυτό είναι ο τρόπος για το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λούκας. Η Επιτροπή μας σαφώς θα επανέλθει στα θέματα αυτά πολλές φορές μάλιστα καθώς θα συζητάμε τους στόχους βιόμιτσιμης ανάπτυξης και καθώς θα διατυπώνουμε θέσεις για τις συμφωνίες αλληλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλο πλαίσιο βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay. Yeah. So we will continue to item... Θα συνεχίσουμε με το θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης που αφορά την κατάσταση στο Μπουρούντι και πιο συγκεκριμένα τη χρηματοδότηση των Μπουρουντιανών στρατευμάτων του ΟΗΕ από το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Παρότι Παρότι δεν προ, περιλαμβάνονται στον προπολογισμό της Ένωσης, ε, τα χρήματα της αναπτυξιακής βοήθειας είναι ευρωπαϊκά χρήματα, επειδή ε, το μέσο αυτό είναι ε, χρη, ε, τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες ΑΚΕ. Και γι' αυτό ακριβώς κινητοποιούνται αυτοί οι πόροι. η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων της και της δημοκρατίας οδηγεί στο να αντιμετωπίζει ακόμα ανθρωπιστική κρίση τον Μπουρούντι. Στην Τανζανία, που είναι η γειτονική χώρα, υπάρχουν περίπου 400.000 πρόσφυγες από τον Μπουρούντι. Για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, έχω τη χαρά να ε, χαιρετήσω τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας ε, Εξωτερικής Δράσης. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Φραντσέσκα Ντιμάουρο καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ναι, ήρθαμε εδώ για να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση στο Μπουρούντι. Όπως γνωρίζετε, το Μπουρούντι είναι ε, σε πολύ εύθραυστη κατάσταση. Υπήρξε πολιτική κρίση και συνεχίζεται από το 2015 με συνεπία της κρίσης αυτής να έχουμε μια οικονομική κρίση και επηρεάζονται και οι χώρες ε, γύρω από τον Μπουρούντι υπήρξε συμπέρασμα του Συμβουλίου από το Μάρτιο του 2016 για την αναστολή ε, της ε, βοήθειας μέσω του ΕΤΑ προς τον Μπουρούντι. Ως όμως άμεση στήριξη προς την κυβέρνηση που αυτό αναστάλει, αναστάλει. Αλλά η στήριξη στον πληθυσμό συνεχίζεται λέει η απόφαση γιατί τη χρειάζεται. Είναι σε δινή θέση ο λαός του Μπουρούντι και θέλουμε να συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε. Αν δείτε και κάποια από τα νούμερα, το 40% του πληθυσμού ε, πλήττεται από ανασφάλεια σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και το 65% ζει ε, σε συνθήκες ε, ακραίας φτώχειας. Κάτι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Το Μάρτιο του 2016 σας είπα, πήραμε αυτή την απόφαση και έκτοτε το ΕΤΑ παίρνει κάποια μέτρα, 55 εκατομμύρια το 2016, 95 εκατομμύρια το 2017 για να καλύψουμε την πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες για τον πληθυσμό, δηλαδή την υγεία, αυτό έχει να κάνει και με τη διατροφή, ασφάλεια τροφίμου, γεωργία και βέβαια πρόσβαση σε βιώσιμη ενέργεια. Είναι σημαντικό επίσης να σημειώσουμε ότι παράλληλα με αυτή τη στήριξη στον πληθυσμό παρέχουμε άμεση υποστήριξη και στην κοινωνία των πολιτών. Για να ξεκολουθήσει να υπάρχει μια κοινωνία των πολιτών, να έχει υποστήριξη και να μπορεί να προωθήσει ε, και να προβάλλει ε, κάποια πράγματα, αλλά και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτό στηρίζει και τους πρασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει ένα έργο, σχέδιο συγκεκριμένο. Εμπιστευτικό, ε, εμπιστευτικότητα, προστασία των ε, υπέρσπιστων ανθρώπων δικαιωμάτων. Μέσω τώρα του ειρηνευτικού μέσου για την Αφρική, African Peace Facility, από το 2015 είμαστε πολύ δραστήριοι και στον τομέα αυτό, με την επέκταση της κρίσης, θέλουμε να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να στηρίξουμε στους παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Αφρικανικής Ένωσης στη χώρα, αλλά και του στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες. Το κάνει αυτό το μέσο το... που σας προανέφερα και ίσως είναι και μια από τις λίγες αποστολές που έχουμε στο Μπουρούντι για να παρακολουθούμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ίσως να το γνωρίζετε, θα μπορούν να το επιβεβαιώσουν και να πούν και άλλα και ή της ΑΕΔ Έχουμε την πολύ καλή συνεργασία Μάλλον υπάρχει το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ που δεν το θέλουν οι Μπουρουντιανοί. Υπάρχει κάποια συζήτηση σε επίπεδο ΟΗΕ, αλλά αρνούνται τις εκθέσεις, ε, απορρίπτουν όλα τα συμπεράσματα του ΟΗΕ, υπάρχει άρνηση. Παρακολούθησα τη κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ δύσκολη. Αλλά αυτό το μέσο μας επιτρέπει να ρίχνουμε μια ματιά ε, και να διαπιστώνουμε ότι δεν είναι καθόλου καλή κατάσταση. Επίση ε, έχουμε την αποστολή Άμισο. Θα θέλετε φαντάζομαι να σα πούμε και για αυτήν την αποστολή. Αν διαβάσετε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαρτίου του 2016 προβλέπετε ότι θα πρέπει να επαναθεωρηθεί, να επανεξεταστεί αυτή η αποστολή, η ειρηνευτική αποστολή στη Σομαλία. Έχει και το Μπουρούντι στρατεύματα στην Άμισο. Και είπαμε ότι πρέπει να το επαναξετάσουμε και να αναθεωρήσουμε την αποστολή αυτή. Γιατί δεν δίνουμε πλέον άμεση υποστήριξη στην κυβέρνηση. Δεν επιτρέπεται. Άρα πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτή την αποστολή και τον τρόπο με τον οποίο στηρίζουμε την άμεση. Άρα τώρα τι έχουμε. Έχουμε ένα μηχανισμό που πηγαίνει στην Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης απευθεία. Εκεί πάνε τα ποσά και αυτοί πληρώνουν τους στρατιώτες. Χρηματοδότηση δηλαδή καμία μέσω των Μπουρουντιανών αρχών. Έτσι έχει κατάσταση. Αυτή είναι η εισαγωγή μου και θα ήθελα να δώσω το λόγο σας, αν έχετε το χρόνο, στους συναντέλφους από την ΕΕ και από το ΕΚΟ. Uh, σας ευχαριστούμε πολύ. Ας ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο της DG ECO, Τόρστεν Μουέντχ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να σας ενημερώσω σύντομα για την κατάσταση των προσφύγων Περίπου 400.000 πρόσφυγες από τον Μπουρούντι βρίσκονται σε όμορες χώρες. Οι περισσότεροι είναι στην Τανζανία, 137.000 είναι εκεί. Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες ζουν σε καταβλισμούς και 100% εξαρτώνται από εξωτερική βοήθεια για να επιβιώσουν. Παράλληλα, το περιφερειακό σχέδιο ανταπόκρισης του 2018 δεν έχει χρηματοδοτηθεί ένα 12% από τα 392 εκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται, ένα 12% μόνο έχει χορηγηθεί μέσω του UNH, μέσω της ΥΠΑ Αρμοστίας για τους πρόσφυγες και επίσης, όπως είπατε, είπατε αυτή η αρμοστία, ενδεχομένως το Μπουρούντι και η προσφυγική κρίση από το Μπουρούντι να γίνει μια ξεχασμένη πλέον κρίση. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2,7 εκατομμύρια έδωσε φέτος σε σχέση με τα 11,7 εκατομμύρια του 2017. Οι πρόσφυγες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιστρέψουν, λέει η επίσημη κυβέρνηση, γιατί έχει αποκατασταθεί πλέον η πολιτική κατάσταση στη χώρα. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως είναι ότι κατά μέσο ώρα έχουμε χίλιους περίπου πρόσφυγες οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα και οι βασικοί λόγοι που έχουν δηλωθεί είναι η ανασφάλεια, ο φόβος και η παρενόχληση. Τώρα να αναφερθώ στην Τανζανία. Ξέρετε ότι παραδοσιακά είναι η χώρα εκείνη η οποία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων από τον Μπουρούντι και αυτό το έχουμε δει εδώ και αρκετό καιρό και μάλιστα βλέπουμε ότι η Τανζανία δεν προτίθεται πλέον να δεχθεί νέους ετούντες άσυλο. Μέχρι πέρυσι πριν Φάτση είχε δώσει αυτόματα το καθεστώς <clears throat> του πρόσφυγα η Τανζανία προς τους πρόσφυγες από τον Μπουρούντι, όμως αυτό έχει σταματήσει. Δεν συμμετέχει πλέον η Τανζανία στο πλαίσιο ανταπόκρισης και αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, στο οποίο προβλεπόντουσαν κάποιες πιο μακροπρόθεσμες λύσεις. Οι αρχές επίση τανζανίε, δεν δίνουν πλέον την υπηκότητα της Τανζανίας για του πρόσφυγες από τον Μπουρούντι, πράγμα το οποίο είχαν κάνει στο παρελθόν και αντίθετα αυτή τη στιγμή ζητούν από τους πρόσφυγες, τους Μπουρουντιανούς, να φύγουν από Τανζανία και να επιστρέψουν στη χώρα τους, χρησιμοποιώντας και αυτή την επιχειρηματολογία που προβάλλει η κυβέρνηση του Μπουρούντι. Και οι δύο χώρες, Τανζανία και Μπουρούντι, συμμετέχουν στην ε, ύπατη αρμοστία και έχουν καταλήξει ήδη από το Σεπτέμβριο του 2017 σε μια τριμερή συμφωνία μεταξύ Μπουρούντι, Τανζανίας και ύπατης αρμοστίας των Εθνών Περίπου 44.000 πρόσφυγες έχουν πάει λοιπόν από την Τανζανία, έχουν επιστρέψει στον Μπουρούντι και συνεχίσει όμως και ασκείται πίεση και από τις δύο πλευρές προκειμένου να επιστρέψουν περισσότεροι Μπουρουντιανοί πρόσφυγες και μάλιστα υπήρχαν και κάποια άρθρα στον τύπο όπου ε, ορισμένοι πολιτικοί από τον Μπουρούντι εκφόβιζαν ορισμένους πρόσφυγες ε, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Μπουρούντι να επιστρέψουν στον Μπουρούντι διαφορετικά κινδυνεύουν με ε, φυλάκιση. Επίσης, βλέπουμε ότι ε, η προσπάθεια αυτή ε, επιστροφής ενός μεγαλύτερου αριθμού προσφύγων από την Τανζανία προ τον Μπουρούντι, ενδεχομένω να μην ευωθωθεί γιατί δεν υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση για έναν τέτοιον ε, επαναπατρισμό. Το πρόβλημα λοιπόν τη χρηματοδότηση δεν έχει να κάνει μόνο με τον επαναπατρισμό, αλλά έχει να κάνει και με τη χρηματοδότηση για την παροχή βασικών υπηρεσιών και στους ίδιους καταβλισμούς. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές περικοπές σε αυτή τη χρηματοδότηση, δεν παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες, περικοπές έχουμε στα προγράμματα επισητισμού, περικοπές επίσης στα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης και αυτό χρησιμοποιείται ως μέθοδος όλο και περισσότερο από τις αρχές Τανζανίας προκειμένου να πιέσουν όλο και περισσότερους πρόσφυγες από τον Μπουρούντι να επιστρέψουν στη χώρα τους. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε βασικές υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τον επισητισμό της, την υγειονομική περίθαλψη. Δεν είμαστε υπέρ της διαδικασίας επαναπατρισμού ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή ασκείται μια ανισό, μια υπερβολική πίεση θα έλεγα στους πρόσφυγες για να επιστρέψουν και δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση η πολιτική στον Μπουρούντι είναι τέτοια ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν περισσότεροι πρόσφυγες. Καταλαβαίνετε ότι οποιοδήποτε επαναπατρισμός, οποιαδήποτε επιστροφή αποφασιστεί θα πρέπει να ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προφανώς θα πρέπει να γίνεται με την ελεύθερη επιλογή των προσφύγων. Δεν μπορούν να καταναγκάζονται σε μια τέτοια απόφαση. Όσον αφορά τώρα την ανθρωπιστική κατάσταση στο Μπουρούντι, για τους εργαζόμενους στα ανθρωπιστικά προγράμματα, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δυσχερής, οι συνθήκες ιδιαίτερα αντίξωες, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί διάβλοι παροχής τέτοιας ανθρωπιστικής βοήθειας η κυβέρνηση, η μάλλον του Μπουρούντι επιτρέπει τέτοια ανθρωπιστική βοήθεια μόνο μετά από φυσικέ καταστροφέ όπω μετά τι πρόσφατε πλημμύρε, αλλά για παράδειγμα δεν επιτρέπεται μια ανεξάρτητη αποτίμηση των ανθρωπιστικών αναγκών, ιδίω στα σύνορα, στην παραμεθόριο δηλαδή με την Τανζανία. Επίση, περιορισμένη δραστηριότητα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων θα πρέπει η δράση του να συνάδει απαραίτητα με τι πρωτοβουλίε και τη βούληση τη κυβέρνηση. Επίσης, υπάρχουν ε, ε, προβλήματα όσον αφορά την ε, ισότητα των δύο φύλων όσον αφορά αυτά τα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Γκεράρντους Γκίλεν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, τώρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στη σημερινή συζήτηση. Εκτιμάμε το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Βουρούντι, που γίνεται μία από τις κρίσεις του κόσμου το που αγνοούμε και το ότι παραμένει στην ημερήσια διάταξη είναι σημαντικό. Από την αναπτυξιακή σκοπιά, η ενίσχυση των προπτικών του πληθυσμού και η βελτίωση της κατάστασης του δικαίου, της ατιμορρησίας και η αποκατάσταση του ε, κράτους δικαίου ε, βοηθούν το πρόγραμμα συνεργασίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη του πληθυσμού του Μπουρούντι είναι, συνεχίζεται. Έχουμε, όπως ακούσατε από τον συνάδελφο, ένα πρόγραμμα 95 εκατομμυρίων, τα οποία ε, έχει εγκριθεί το 2017. Μας ε, ανησυχούν οι παραβιάσεις των Ευρωπαίων δικαιωμάτων που δημοσίευσε στην έκθεσή της ε, η Επιτροπή Έρευνες το Σεπτέμβριο. η τα μέλη της Επιτροπής Έρευνας δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτα στο Μπουρούντι. Ε, απαιτείται ε, το Μπουρούντι να ανοίξει το, διάλογο με, με οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στηρίζουμε την παράταση της εντολής της Επιτροπής Έρευνας και ε, υπάρχει και ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επ' αυτού ο σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων πιστεύουμε ότι δημιουργεί στη δημιουργία, ε, συνεισφέρει στη δημιουργία ευημερούσας και σταθερής κοινωνίας. Και είναι σημαντικό για τον Μπουρούντι. Είμαστε πεπισμένοι ότι ένας διάλογος μεταξύ των, ε, των Μπουρουντιανών είναι ο τρόπος για να προχωρήσουμε και τον Οκτώβριο θα γίνει μια επόμενη συνεδρίαση που μπορεί να αποβεί σημαντική για την ιστορία της χώρας. Έτσι ενθαρρύνουμε όλους τους παράγοντες να συμμετάσχουν ενεργά ε, στο διάλογο αυτό και στις εκλογές ε, που θα γίνουν το 2020. Η διευκόλυνση του διαλόγου στο εσωτερικό της χώρας ε, μέσω της Αφρικανικής Ένωσης δείχνει ότι η διαμεσολάβηση της περιοχής είναι σημαντική. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει στενή συνεργασία με τέρους όπως την κοινότητα Ανατολικής Αφρικής, την ε, και το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών. Και θα σταματήσω στο σημείο αυτό. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Υπάρχουν σύντομες παρατηρήσεις ή σχόλια. Ο κύριος Τσέλερ. Ευχαριστώ. Ε, Πραγματικά είναι πάρα πολύ σχετική η κατάσταση. Το καθεστώς κάνει δικτατορικό μόνο μπορεί κανείς να το ε, περιγράψει και σίγουρα ε, θα πρέπει να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια, ιδίως ό,τι αφορά τους πρόσφυγες στην Τανζανία και στις άλλες γειτονικέ χώρες. Το είπατε κι εσείς όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει κανεί στη χώρα. Με ποιον τότε ε, συνεργαζόμαστε εκεί, αν θέλουμε να δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή. αποκλείεται οποιαδήποτε συνεργασία με την κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, οι οργανώσει κοινωνία των πολιτών εκεί πέρα είναι απαγορευμένε. Σε ό,τι αφορά την Άμισον και τα μπουρντιανά στρατεύματα, είναι ένα μέσο καταστολής ο στρατός. Το καθεστώ ε, του Κουρουσί Κάνια. και υπάρχουν ε, ακριβά, ακριβές αμοιβέ για τους στρατιώτες. Το African Peace Facility νομίζω ότι παίρνει ε, το 90% από το ΕΤΑ. Επίσης ακούμε για τα μπορουντιανά στρατεύματα ότι δεν είναι και τόσο αξιόπιστα και σομαλικές περιοχές που πρέπει να προστατεύουν τον άμαχο πληθυσμό δεν το πράττουν. Και με την Al-Shabaab ε, δημιουργήθηκε ένας ευρύτερος τελικά κύκλος ε, τρομοκρατίας. Τι επιπτώσεις είναι αυτές, ε, τι συμπεράσματα αντλούμε από όλες αυτές τις επιπτώσεις. Η κυρία Χόιμπουχ. Yeah, Σας ευχαριστώ. Πολλά μας είπατε για την κατάσταση το Μπουρούντι. Ο τίτλος όμως είναι και χρηματοδότηση των Βρυτανών στρατευμάτων από το ΕΤΑ και το Άφρικα που Facility. Δεν είπατε τίποτα γι' αυτό, ούτε κανείς από τους τρεις. Το είπε και ο προλαλής σας το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό. Υπάρχουν χρήματα για τις αμοιβέ των στρατιωτών που βγαίνουν από αυτό το μέσο. Είναι τεράστια τα ποσά. Υπάρχουν διαψεύσεις, αλλά τον Ιούνιο του 2017 ένας εκπρόσωπος ε, του στρατού στο ε, γαλλικό ραδιόφωνο είπε διαφορετικά πράγματα. Τι γίνεται με τα χρήματα αυτά. Υπάρχει και μια τράπεζα για τους στρατιώτες που έχουν τους, τους λογαριασμούς τους. Το ξέρετε αυτό. Η Κομισιόν το ξέρει. Το λέτε με την Αφρικανική Ένωση. Υπάρχει συντονισμό ε, του μέσου στήριξη από την Ευρωπαϊκή Αφρικανική Ένωση. Από αυτά τα περιστατικά έχουν αντληθεί διδάγματα. Και επειδή τώρα διαπραγματευόμαστε το πολιτές δημοσιονομικό και θα υπάρχει αυτό το μέσο διευκόλυνσης. Πώς θα το αντιμετωπίσετε, υπάρχουν κάποια προληπτικά μέτρα για να μην ξαναγίνει στο μέλλον κάτι αντίστοιχο. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. I will ask short uh, answers. Answers. Παρακαλώ σύντομες απαντήσεις. Ποιος θέλει να απαντήσει. Ένα λεπτό έχετε με ποιον συνεργαζόμαστε στον Μπουρούντι. Είναι 1,9 εκατομμύρια το ποσό της ανθρωπιστικής βοήθειας στον Μπουρούντι. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού είναι ο φορέας με τον οποίο συνεργόμαστε. Έχει πρόσβαση μέχρι τις φυλακές. Αυτό στον τομέα της προστασίας. Και υπάρχει ένα μικρό ποσό για το συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας, ε, το ΟΤΣΑ, το γραφείο αυτό, που δίνει advocacy και συντονισμό μικρά προγράμματα. Υπάρχει και ε, εθελοντισμός από Ιταλία, υπάρχουν και κάποια σχέδια ε, για τη διατροφή των παιδιών και έπειτα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση έχουμε κάποιες διαπραγματεύσεις για όσους επιστρέφουν στη χώρα να έχουν προστασία ε, δηλαδή και να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει με τους, ε, πανα, τους παλινοστούντες τέλος πάντων να δούμε πώς έχει κατάσταση μετά από 6-8 χρόνια. Αυτό το κάνουμε σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση. Με αυτές τις οργανώσεις ουσιαστικά συνεργαζόμαστε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και Μούνιχ. Άλλα σχόλια υπάρχουν. Ναι. Εγώ, πολύ σύντομα. Για τον τίτλο, ναι, πράγματι. Αυτό αφορούσε, θεωρούσα την Αφρικανική Ένωση πιο πολύ, για το ΝΟΙΑ δεν μπορώ να πω, γιατί αυτοί οργανώνουν ε, τις ενευτικές αυτές αποστολές και εμείς δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, ε, τα κράτη-μέλη. Για το EPF, το μέσο στήριξης δηλαδή και για τα πορδιανά στρατιώτα που δεν είναι αξιόπιστα και δεν ε, κάνουν αυτά που πρέπει. Ε, δεν ξέρω ε, αν έχετε διαβάσει την εκτισάμιση, αλλά δεν λέει τίποτα για κακή συμπεριφορά αυτών των στρατιωτών. Δεν έχουμε στοιχεία για το κατά πόσον υπάρχει αυτή η μεταφορά των πιστώσεων. Εμεί έχουμε μια σύμβαση με την Επιτροπή Αφρικανικής Ένωσης και κάναμε και μία, με έναν έλεγχο για να που πάνε τα λεφτά. Και τα προκριτρακτικά αποτελέσματα, δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχο, δείχνει ότι τα κονδύλια εμεί που δίνουμε στην Επιτροπή Αφρικανική Ενότητα πάνε πράγματι ε, σε ε, έναν λογαριασμό ε, που είναι όμως λογαριασμός των στρατιωτών, παίρνει το 100%. Τώρα τίποτα άλλο δεν ξέρω. Κάποιες καταγγελίες υπάρχουν, αλλά δεν βλέπουμε στον έλεγχο αυτούς, ε, αυτές τις ροές. Και για το επόμενο πολιετές, ναι, υπάρχει πρόταση για το νέο African Peace Facility ή μάλλον Peace Facility, που δεν θα, δεν θα περιορίζεται δηλαδή μόνο στην Αφρική. Και οι συζητήσεις ακόμη συνεχίζονται και φαντάζομαι ότι τα θέματα αυτά μπορούμε να τα ξαναθέσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε εκ του τη γενική κατάσταση στο Μπουρούντι. και το τι θα αποφασιστεί σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και τη δράσεις του ΟΗΕ. Thank you very Ξελίσσονται άλλωστε τα πράγματα τάχιστα. Πάμε στο 11. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τι τροπολογίες του σχεδίου έκθεση για την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα τη εκπαίδευση. Θα θυμάστε ίσως ότι είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων από το σχεδίο εκθέσεως αυτού στις 12 Ιουλίου. 120 τροπολογίες έχουν κατατεθεί. I will now give the floor to Vincent Θα δώσω το λόγο στον Βενσάν Pellon για να μας δώσει τα δικά του σχόλια για τις τροπολογίες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε δίκιο, κυρία Πρόεδρε. Όντως, 120 είναι τροπολογίες που κατατέθησαν. Πρέπει να πω ότι είχα πει ότι δεν θα πρέπει να αλλοιώσουμε σε καμία περίπτωση τους βασικούς άξονες της έκθεσης, να έχουμε μια συμπαγή έκθεση. Νομίζω ότι το καταφέρουμε αυτό, διότι από τις 120 αυτές τροπολογίες νομίζω ότι μπορούμε μέσω του συμβασμού να συμπεριλάβουμε τα δύο τρίτα αυτών των τροπολογιών και μπορώ να πω ότι κάποιες τροπολογίες όντως επιφέρουν εύχριστες διευκρινήσεις. Ευχαριστώ τους συναδέλφους οι οποίοι απουσιάζουν όμως όσον αφορά το ψηφιακό περιβάλλον, όσον αφορά την ισότητα των φύλων, όσον αφορά την πολιτική χωρίς αποκλεισμούς. Πολλές τροπολογίες είχαν να κάνουν με τις επίγουσες καταστάσεις, με την κατάρτιση των δασκόντων, και κάτι το οποίο είχαμε καλύψει και κάτι τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων, τη διασύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την υγεία. Νομίζω ότι οι περισσότερες δυσκολίες έχουν να κάνουν ίσως με εθνικές νοοτροπίες και στάσεις εδώ πέρα όσον αφορά την κρατική ενίσχυση, τις δημόσιες ενισχύσεις και επιδοτήσεις όσον αφορά τα συστήματα εκπαίδευσης. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε εδώ πέρα όλοι τις ίδιες εμπειρίες, τη ίδια Στόχος μου σε καμία περίπτωση δεν ήταν να περιορίσω την ελευθερία επιλογών, αλλά να διασφαλίσουμε ότι στο νέο αυτό σύστημα όλοι οι μηχανισμοί οι οποίοι θα προβλέπονται να μπορούν αν μη τι άλλο κάπως και κάπου να ελέγχονται. Ξέρετε ότι εδώ πέρα αυτό που μας ενδιέφερε είναι ότι πέρα από τους δημόσιους πόρους θέλαμε να έχουμε και ένα σημαντικό επίπεδο απόδοσης των επενδύσεων. Ξέρετε ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε πολλές φορές ακόμα και κάποιες επενδύσεις για τις οποίες δεν θα προβλέπεται αναγκαστικά μια απόδοση. Προσπαθήσαμε πάντως για τις περισσότερες τροπολογίες να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή διατύπωση. Ήρθα σε επαφή και με τους σκιώδεις συγητές, γιατί είδα ουσιαστικά ότι ε, όλοι προασπίζαμε τους ίδιους στόχους, αλλά πολλές φορές ακολουθούσαμε διαφορετική διατύπωση. Επίσης είδαμε ότι πολλές φορές υπάρχουν κράτη εποφελούμενα από τα προγράμματα αυτά τα οποία δεν μπορούν από μόνα τους να οργανώσουν τους ελέγχους αυτούς. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αναφερόμενος τουλάχιστον στη δικιά μου τη χώρα, τη Γαλλία, η Γαλλική Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας ντρέπεται ουσιαστικά να δίνει δημόσιους πόρους σε έναν διεθνή ιδιωτικό οργανισμό που ουσιαστικά κάνει την εκπαίδευση, την προωθεί την εκπαίδευση σαν να ήταν ε, εμπόρευμα και πολύ συχνά αυτό γίνεται μάλιστα σε φορολογικούς παραδείσους. Ξέρετε ότι ε, υπάρχουν ε, και διαφημίσεις όσον αφορά <clears throat> επενδύσεις που θα μπορούσαν να δώσουν ακόμα και μια απόδοση της τάξης του 20% σε ορισμένες αφρικανικές χώρες. Ιδιωτικά ταμεία τα οποία μέσω διαφημίσεων προωθούσαν τέτοιες επενδύσεις. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν μπορούμε μέσω της βασικής εκπαίδευσης να επιτρέπουμε σε κάποιους να κερδοφορούν. Ιδίω όταν αναφερόμαστε σε μαθητές και σε παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση έσχατης φτώχειας. Νομίζω πάντως ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε συμβασμούς. Μέχρι την Τετάρτη θα είμαι σε θέση, θα να προτείνω συμβαστικές προτάσεις στους σκιώδεις ηγητές. Θα ψηφίσουμε στις 9 Οκτωβρίου. Θα πρέπει ή θα ήταν καλό σκόπιμο να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού συνεδριάσει στις αρχές Δεκεμβρίου η ε, ομάδα της Παγκόσμιας Εταιρικής Σχέσης για ε, την εκπαίδευση. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και με τους όρους που χρησιμοποιούμε. Καλή κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, αλλά από την άλλη οι ιδιωτικέ επιχειρήσεις δεν είναι συνώνυμο των, ε, της κοινωνίας των πολιτών και δυστυχώς σε ορισμένες τροπολογίες υπήρχε μια σύγχυση ανάμεσα στους δύο αυτούς όρους. Συνεχίζεται η εργασία, είμαι αισιόδοξο, θα καταλήξουμε πιστεύω σε 23 συμβαστικέ προτάσει, οι οποίε θα καλύψουν πιστεύω τα δύο τρίτα των τροπολογιών. Ενδεχομένω να έχουμε και κάποιες επιπλέον τροπολογίες οι οποίες θα μπορούσαν να εγκριθούν πέρα από τις συμβαστικές τροπολογίες. Το πιο σημαντικό να καταφέρουμε όλοι να επικεντρωθούμε σε κάποιες βασικές προτεραιότητες. Αυτές ακριβώς θα πρέπει να προωθούμε μέσω της έκθεσης αυτής, προκειμένου η έκθεση αυτή να μπορεί να βαρύνει ενώπιον των υπολείπων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, κύριε Πεϊόν δουλέψατε πολύ σκληρά και χειριστήκατε πολύ καλά αυτές τις 120 τροπολογίες να μας, και για να μας παρουσιάσετε το πακέτο αυτό. Η ψηφοφορία, όπως ε, είπατε, θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή είναι πεντασέλιδη και ε, καλύπτει ολόκληρο το πακέτο με το οποίο, ε, ε, το οποίο μας απασχολεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω να ε, θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, έχω χρόνος ερωτήσεων. Δεν έχουν ληφθεί ερωτήσεις για την συνεδρίαση αυτή. Τα διάφορα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που έχει κάτι να προσθέσει στα διάφορα. Όχι. Οπότε έχουμε να ορίσουμε την επόμενη συνεδρίασή μας, η οποία θα γίνει στις 8 και 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις ώρες που το πρόγραμμα που βλέπετε στην ημερήσια διάταξη, στο σημείο αυτό, ολοκλήρωσε, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής ΔΕΒΕΣ. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.